yes, I'll speak in English. Okay, good. Mesdames, Messieurs, bonjour. Allez, nous commençons notre séance. L'audition par la jeunesse d'aujourd'hui est diffusée sur le web. Η σημερινή ακρόαση θα διαδοθεί, θα αναμεταδοθεί, με συγχωρείτε, στο ίντερνετ. Είναι ένα α, α, από μία από τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρώπης για τους νέους. Λοιπόν, οι νέοι ολόκληροι της Ευρώπης μας παρακολουθούν. Μπορείτε λοιπόν να τους χαμογελάσετε. Καλείστε να συμμετέχετε και στη συζήτηση επιγραμμικά, γιατί και εμείς χρησιμοποιούμε hashtag. Οπότε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, βάζετε hashtag ε, ε, ε ε, 2018 θα το δείτε και στην οθόνη εδώ εντό τη αίθουσα. Όπω γνωρίζετε, το Ευρωκοινοβούλιο διοργανώνει το Κοινοβούλιο τη Νεότητα από το 2014. Φέτο είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή 9.000 νέων, όπου ορισμένοι ευρωβουλευτέ έκαναν ε, μεγάλη επιτυχία. Ε, έκαναν ένα σλάμ ε, και εγώ μαζί ε, δηλαδή έγινε ένας διαγωνισμός ανάμεσα σε διάφορους ε, ράπερ και εγώ ήμουν εκεί και πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν είδα σε ποιο βαθμό η συζήτηση και οι ιδέες ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, θετικές και μάλιστα στραμμένες προς το μέλλον. Οι ε, ναι, νέοι λοιπόν μπορούν να σημάνουν τη διαφορά. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η συμβολή τους ε, πρέπει και μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ατζέντα του Κοινοβουλίου και ε, ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον έτσι να πάμε σε μια δημοκρατία πολύ πιο ευρωπαϊκή και πιο δυναμική. Αυτό χρειαζόμαστε στην Ευρώπη σήμερα. Για να καθησυχάσουμε, για να εξασφαλίσουμε μάλλον αυτό, την πολιτική συνέχεια όλων αυτών των εκδηλώσεων, το Προεδρείο αποφάσισε ότι στη συνέχεια αυτών των εκδηλώσεων θα έπρεπε να γίνει συζήτηση εντός των θεσμών μας στις επιτροπές που είναι αρμόδιες. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Άρα λοιπόν στόχος αυτής της ανταλλαγής απόψεων και στρέφομαι και προς εσάς και σας κοιτώ γιατί θα σας ακούσουμε για να δούμε εάν οι προτάσεις σας για το μέλλον της νεότητας ε, ε, δεν θέλουμε μόνο να σας ακούσουμε, θέλουμε και να συζητήσουμε μαζί σας για να δούμε και να ακούσουμε τι περιμένετε εσείς από τους ε, εκπροσώπους σας και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μετά από αυτή την τρίτη λοιπόν έκδοση, εκδοχή, θέλουμε να σας υποδεχτούμε. Είναι τρεις συμμετέχοντες, πιστεύω πως θα μας κάνουν να ονειρευτούμε. Προσπαθώ να σας πιέσω, λέει η Πρόεδρος, να ακούσουμε τις ανησυχίες σας, τις προσδοκίες σας και θα χρειαστεί και να μας πείσετε. Δεν αρκεί να έχετε λοιπόν τις καλές ιδέες, πρέπει και να μας πείσετε για τα θέματα που μας αφορούν εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα μας μιλήσετε για τις ιδέες σας, τις στρατηγικές σας για να προωθήσουμε μια νέα κινητικότητα αύριο μεθαύριο και τον τουρισμό με τρόπο καινοτόμο και βιώσιμο. Ξέρετε ότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Είναι προτεραιότητά σας, δεν είστε βέβαιοι μάλιστα. Μια κινητικότητα λοιπόν που να είναι και ε, προσιτή σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τρεις νέους ομιλητές που θα μας δώσουν ιδέες και εμείς οι ευρωβουλευτές θα ε, είμαστε οι δέκτες αυτών των ιδεών. Είστε ευπρόσδεκτοι λοιπόν εδώ και σας τους παρουσιάζω αμέσως. Φιλίπ Βος. Ε, είστε 29 ετών και είστε Γερμανός. Μάλιστα, πολύ ωραία. C'est vrai. Πελομή Φαντάρ. Πελομή Φαντάρ. Φανταρέ. Μάλιστα. Εντάξει, στα γαλλικά θα διαβαζόταν Φαντάρ. Είστε 23 ετών, είναι πιο νέα από εσά. Βλέπετε και εσείς είστε Ισπανίδα, Νιγηριανής προέλευσης. Η Εύα Γκούντερ, εσείς είστε ακόμα πιο νέα, 22 ετών μόλις και είστε και εσείς Γερμανίδα. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, λοιπόν, και στο όνομα αυτής της Επιτροπής σας καλωσορίζω και δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο σε αυτή μας την ακρόαση, αλλά καθένας θα πάρτε το λόγο για δύο λεπτά και μετά θα δώσουμε το λόγο στους διάφορους ε, βουλευτές που θα έρθουν ε, για να δούμε λοιπόν και εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά. Φιλίπ, εγώ ξεκινάμε με εσά. Βάζω εδώ χρονόμετρο. Είστε έτοιμος? C'est bon <laughs> Allez, on y va. Thanks, Karine. Uh, thanks for having us. Um, Ευχαριστώ, Καρίμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, αυτό που με απογοητεύει είναι ότι έχω ένα πλαστικό μπουκάλι μια χρήση μπροστά μου, αλλά τέλο πάντων δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Το πρώτο θέμα είναι οι ε, εκπομπέ άνθρακα και πώ ε, θα μπουν στο σύστημα ETS. Γιατί οι πολλέ εκπομπέ του άνθρακα είναι από τα βασικά προβλήματα στον τομέα του μεταφορά και του τουρισμού. Οι εκπομπέ ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τα πρότυπα εκπομπών. Ο κανονισμό είναι σημαντικός ε, που τα διέπει όλα αυτά, αλλά δεν φτάνει. Για να περιορίσουμε δραματικά τα αέρια του θερμοκηπίου και να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα στις μεταφορέ μέχρι το 2050, χρειαζόμαστε περισσότερες ενέργειες. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο τομέα των μεταφορών στο EUTS e και θα πρέπει να γίνει ήμια ανοιχτό το σύστημα. Το EU ETS είναι τεχνολογικά ουδέτερο και αποτελεσματικό μέσο γιατί οι περικοπές, οι μειώσει γίνονται εκεί που αυτό είναι φθηνότερο. Μπορεί να επηρεάσει το, όλο το φάσμα των ε, ε, μειώσεων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και με τη βελτίωση ε, της συμπεριφοράς ε, των οδηγών και το καθεξής, πώς θα συμπεριληφθεί ο κλάδος στο EU ETS. Πρέπει να ρυθμίζεται ανάντι ο κλάδος, σε επίπεδο δηλαδή των παρόχων ε, καυσίμων και έτσι μπορεί να περάσει όλο αυτό ε, στους ε, καταναλωτές και η κατανομή να μην γίνεται δωρεάν, αλλά με βάση δημοπρασία. Το ίμιο ανοιχτό σύστημα σημαίνει ότι θα, οι μειώσει θα γίνουν στον τομέα των μεταφορών και όχι σε άλλους και περιορίζει ε, και εμποδίζει την εξαγορά πιστοποιητικών από, από άλλους κλάδους και έτσι είναι πιο δίκαιο το σύστημα. Το EU ETS μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές και να δημιουργήσει κίνητρα για επιχειρήσεις για να έχουν βιώσιμες τεχνολογίες. Αυτό χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας και του βιωτικού επίπεδου στις ευρωπαϊκές πόλεις. Merci beaucoup, Philippe. Ευχαριστούμε πολύ, Φίλιπ Βος, για την παρέμβασή σας. Δύο λεπτά τώρα έχει η Εύα Γκούντερ. Παρακαλώ. Thank you. Um, I'll speak in German. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γερμανικά. <laughs> Die Idee, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist zwar idealistisch. Σήμερα μπορεί να σας παρουσιάζω κάτι που ακούγεται ιδεαλιστικό, αλλά είναι εφικτό δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες στις ευρωπαϊκές πόλεις. Στο European Youth Event δεν υπήρχε επαρκής ε, αναφορά σε άλλες ζητήματα όσο στις δημόσιες δωρεάν συγκοινωνίες. Είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει όλους. Κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις ήδη το έχουν κατανοήσει. Η Εστονία είναι προς το παρόν το καλύτερο παράδειγμα αλλά και σε άλλες ε, χώρες υπάρχουν ε, εκπτώσεις για τους φοιτητές, για παράδειγμα. Αλλά τι γίνεται με τον απλό εργαζόμενο. Οι δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες ήταν ένα σημαντικό μέτρο ε, για να καταπολεμήσουμε τον καταγερματισμό. Μετά και υπάρχει μια οικολογική διάσταση αν μειώσουμε τον αριθμό των αυτοκινήτων ε, στους ε, δρόμους, θα είχαμε περισσότερο χώρο για τα ποδήλατα και θα ήταν ε, λιγότερο επικίνδυνη ζωή για τους ποδηλάτες. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα για την υλοποίηση είναι ένα σχέδιο δράσης. Υπό το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε ως στόχο τις δωρεάν δημόσιες ε, συγκοινωνίες ε, στις ε, πόλεις με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο Ταλίν, για να χρηματοδοτηθεί αυτό το project, χρησιμοποιούνται οι φόροι εισοδήματος. Και μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και άλλες πόλεις. Και εφόσον λένε και περισσότεροι ε, μετακομίζουν προς τα αστικά κέντρα, αυτό θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Φίλιπ Βος. Α, ναι, να σας εξηγήσω. Ο κάθε ομιλητής θα πάρει το λόγο δύο φορές. Για να δώσει δύο ιδέες. Δηλαδή, μετά Φιλίππε, δεν θα, δεν θα μιλήσεις άλλο. Ναι, κατάλαβα. Η δεύτερη μου ιδέα αφορά την εισαγωγή εφιών δημόσιων ποδηλάτων η κοινή χρήση ποδηλάτων και αυτοκινήτων αυξάνεται, ωστόσο ακόμα κυριαρχούν τα γεωταχή στις, στην κυκλοφορία στις πόλεις. Ε, προκαλούν ε, ρήπανση του αέρα, παίρνουν χώρο. Τα ευφυή λοιπόν ποδήλατα είναι μια εναλλακτική. Στην ουσία πρόκειται για ηλεκτρικά ποδήλατα που μπορούν να αποθηκεύσουν την ενέργεια που παράγεται ενώ κανείς κάνει πετάλι και την χρησιμοποιούν όταν ε, βρεθούν σε ανηφόρα. Δεν χρειάζεται δε, να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο γιατί φορτίζουν όσο ε, κανείς ε, τα χρησιμοποιεί. Τώρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ε, κοινή χρήση αυτών είναι πολύ καλύτερα από τα συμβατικά αυτοκίνητα. Τώρα, για να αυξηθεί ο αριθμός των κοινή χρήσης ποδηλάτων θα πρέπει να αυξήσουμε την απομάκρυση, την, ε, την κατάργηση της χρήσης του άνθρακα από τις δημόσιες μεταφορές, να αυξήσουμε τις ε, λωρίδες, τις ειδικέ ε, για τα ποδήλατα και έπειτα να συνδέσουμε μεταξύ τους και τις πόλεις ώστε να ακολουθήσουμε τις πόλεις που έχουν πρωτοπορήσει στη υποδηλασία όπως η Κοπεχάγη. Να συντονιστούν επίσης ε, τα σήματα κυκλοφορίας και τα φανάρια, ειδικά στις ώρες εχμής είναι μια καλή εναλλακτική στα αυτοκίνητα. Εάν χρησιμοποιήσουμε τα FEE ποδήλατα θα βελτιωθεί και δραστικά η ποιότητα του αέρα και ίσως να φτάσουμε και γρηγορότερα τους ενεργειακούς στόχους στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή σας την παρέμβαση και τις ιδέες σας και τώρα θα το συζητήσουμε αμέσως αυτή την ιδέα με τον Βιν Βαντερκάμπ που είναι μέλος της ομάδας του ΕΛΚ και συντονιστής στην ομάδα μας. Έχεις το λόγο, Βήμα σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Παρακολούθησα την... Και εγώ θα μιλήσω τη μητρική μου. Περιμένω να φορέσετε όλοι τα ακουστικά σας. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ αυτούς τους τρεις σκεπτόμενους νέους. Και εμείς Ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρόμαστε που βλέπουμε πραγματικού ανθρώπους με πραγματικέ ιδέες που δεν ε, ζουν μέσα στη φούσκα που ζούμε εμεί. Προς τον Φίλιπ Βό, ένα ερώτημα. Είστε συγγενείς του Άξελ ή Είναι συνονο... Είστε απλά συνανόματοι. Έχουμε έναν συνάδελφο που λέγεται Άξελ Βό και είναι από τη Βόνη. Τέλο πάντων. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι γιατί θέλετε συνεχώς να τιμωρείτε. Δεν είναι καλύτερα να πούμε ότι ας πούμε στο κέντρο μιας πόλης δεν θέλουμε ε, μηχανές ε, θέλουμε ηλεκτρικά οχήματα. Γιατί εσείς θέλετε ποινές και κυρώσεις ότι πρέπει να μπούμε στο ευρωπαϊκό ETS. Ε, ε Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απλώς χρειάζονται ε, το όχημά τους, μεταφορείς, ο φούρναρης της γειτονιάς. Γιατί να τους τιμωρήσουμε. Δεύτερον, το ζήτημα των συνόρων. Όσοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα απογίνουν. Οι πολίτες της Σερβίας που πηγαίνουν στην Ουγγαρία. Οι Ουκρανοί που έρχονται στην Πολωνία αυτοί μπορούν να οδηγήσουν ελεύθερα. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Και ένα ερώτημα προς την Εύα. Εγώ βέβαια προέρχομαι από ένα συντηρητικό κόμμα. Το θεωρώ εξαιρετική ιδέα. Αλλά ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Ο φορολογούμενος. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το τίμημα και με κάθε ειλικρινία βλέπω ότι υπάρχουν πόλεις στην Ευρώπη που ήδη έχουν εφαρμόσει την ιδέα σου και εσύ ανέφερες ε, το Ταλίν. Για κάποιες ε, πόλεις είναι καλύτερο να δίνουν ε, δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες παρά να έχουν ρήπανση σε όλη την πόλη με, τα, με τις μηχανές καύσης. Αλλά με προβληματίζει λίγο αυτό. Ο Φιλίπ θέλει να τιμωρεί και η Εύα λέει ότι όλα πρέπει να δίνονται τζάμπα. Εμένα με δυσκολεύουν αυτές οι δύο ιδέες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αγωγούνταλόν. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μας για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή. Παρατηρώ ότι οι τρεις πρώτες ε, παρεμβάσεις σας αφορούν τη σημασία και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι δημόσιε συγκοινωνίε, οι μεταφορέ μάλλον ευρύτερα, ε, για το μέλλον μα και πώ μπορούμε να έχουμε περισσότερη κινητικότητα. Εμεί αυτό έτσι κι αλλιώ ε, προασπίζουμε σε αυτή την Επιτροπή, αλλά θέλουμε μια κινητικότητα παράλληλα που θα προστατεύει περισσότερο το περιβάλλον, τον αέρα που αναπνέουμε και θα είναι και πιο προσβάσιμη, γιατί σήμερα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί πολύ σε αυτή την Επιτροπή είναι ο γεωγραφικός ε, κατακαιρματισμός. Υπάρχουν δηλαδή εκείνοι που εύκολα ε, μεταφέρονται, έχουν πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες ε, που είναι εύκολα προσβάσιμες και οικονομικές και υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Και συχνά εκείνοι ρηπαίνουν περισσότερο γιατί πρόκειται για παλαιά οχήματα. Είναι μια συζήτηση που έχει προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία, αν το έχετε δει. Και σας υπενθυμίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις, όχι μόνο η Γάλλοι, αλλά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, για να κινηθούμε προς μία πιο καθαρή, αλλά και πιο προσβάσιμη κινητικότητα. Πώς λοιπόν θα εφαρμόσουμε προτάσεις είτε όπως αυτή για το ETS είτε όπως αυτή για τις δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες και μετά τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Όλα αυτά θα πρέπει κάπως να τα συγκεράσουμε. Και στις προτάσεις ε, που υποβάλλατε θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ο δωρεάν χαρακτήρας ε, θα αφορά κυρίως τις πόλεις και μάλιστα τις πλούσιες πόλεις. Γιατί ε, ε, θα πρέπει να υπάρχουν δημοτικοί φόροι που θα καλύπτουν αυτά που αυτή τη στιγμή καλύπτονται με τα κόμιστρα. Αλλού όμως δεν θα μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Υπάρχουν ε, και άλλοι τρόποι να περιορίσουμε το κόστος των δημοσίων συγκοινωνιών. Ο ΦΠΑ, αν έπεφτε ο ΦΠΑ στο 5% στις δημόσιες συγκοινωνίες, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο, φθην... να δημόσιες συγκοινωνίες. Γιατί το θέμα των μεταφορών δεν είναι μόνο εμείς που ε, μετακινούμαστε, αλλά αφορά και τους εργαζομένους του κλάδου. Σας ενδιαφέρει εσάς η κατάσταση των εργαζομένων του κλάδου των μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και για αυτές τις παρεμβάσεις. Ε, συγχαρητήρια που βρίσκεστε εδώ. Βεβαίω η κοινωνική διάσταση είναι σημαντική και η κινητικότητα, αλλά σημαντικότερο από την κινητικότητα είναι η διατροφή. Και πάρα πολλά παιδιά στην Ευρώπη ε, δεν ε, έχουν ε, να φάνε. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει δωρεάν διατροφή για όλου. Και όσο δεν υπάρχει αυτό, εγώ πρέπει να σα πω ότι είμαι λιγάκι επιφυλακτικό στο να υπάρχουν δωρεάν μετακίνησει. Όμω θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κοινωνικά και οικονομικά πιο αδύναμοι. Στο Βερολίνο, παραδείγματο εδώ και 25 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί ε, τα τέλη για την ε, στάθμευση. Ε, και αυτό το θεωρώ ότι είναι κάτι απαραίτητο. Στη Γερμανία κάθε χρόνο έχουμε 50 εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται σε διάφορες ενέργειες που όμως βλάπτουν το περιβάλλον. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι και πράσινο, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όσον αφορά τις ε, μετακινήσεις της πόλης, ομολογώ ότι το θέμα δεν είναι να έχουμε και άλλο αυτοκίνητο. Ο Hans jurgen Vogel το 1972 ήταν πάρα πολύ νέος, δήμαρχος τότε στο Μόναχο και είχε πει ήδη πριν από 46 χρόνια ένας σοσιαλδημοκράτης ότι το αυτοκίνητο δολοφονεί της πόλη μας. Αν λοιπόν όλα τα αυτοκίνητα είναι πια ηλεκτρικά, ε, τότε πράγματι θα προχωρήσουν οι πόλεις. Απέχουμε βέβαια από αυτό, άρα πρέπει να επενδύσουμε εκεί όπου μπορούμε τις πόλεις να τις κάνουμε καλύτερα βιώσιμες για τους ανθρώπους και όχι για τις ε, ίδιες τις πόλεις. Ε, το θέμα με τα ποδήλατα είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά τα ηλεκτρικά ποδήλατα και ακόμα και ο Γερμανός ε, υπουργό Μεταφορών έχει αποφασίσει να προχωρήσει αυτό το θέμα των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για σκεφτείτε, Βερολίνο, ε, Παρίσι, ε, Μόναχο και Μαντρίδη θα έχουν εξαφανιστεί ή έχουν ήδη εξαφανιστεί το 60% των αυτοκινήτων και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν εγγύησει. Εκεί πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε. Εγώ δεν θέλω να έχουμε δωρεάν αστικές μεταφορές. Εγώ μπορώ να το πληρώνω. Εκείνοι όμως που το χρειάζονται, αυτοί ε, επιδοτούνται με 40 ευρώ για τις μεταφορές, αλλά χρειάζονται περισσότερα χρήματα πράγματα, γιατί στο Βερολίνο είμαστε διπλά πιο ακριβοί από ό,τι παραδείγματο χάνει σε άλλες πόλεις. Ως εκ τούτου να ακολουθήσουμε την εξή κατεύθυνση. Ναι, μεν χαμηλότερα εισιτήρια, αλλά οι εισοδηματικά και κοινωνικά δύναμη να στηρίζονται και όχι μόνο κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατιών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κράμερ. Εν συντομία και εγώ επειδή έβαλα το, όνομά μου στον κατάλογο μελητών, Φιλίπ, συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει κάπως να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας, ιδίω ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Ένα πλανήτη έχουμε μόνο και οι μεταφορές είναι ένας από τους κλάδους ε, που ρηπαίνουν περισσότερο με πολλά αέρα του θερμοκηπίου εδώ και 30 χρόνια. Ε, βέβαια το έχουμε κάνει πλέον μια πολύ σημαντική ε, προτεραιότητα. Τώρα, για τους φόρους που ανέφερες. Εμείς την έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, υπάρχει το ευρωπαϊκό τέλος που ψήφισε η Ευρωπαϊκή, η δική μας μάλλον Επιτροπή. Η κυρία Γανόντα Βον, είπε ότι τα πρέπει τα φορτηγά να ε, φορολογούνται και να μην βρίσκουμε πλέον ε, εμπορεύματα στα φορτηγά, αλλά στα τρένα, για παράδειγμα. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά στο σύστημα ETS και τα λοιπά, θα πρέπει να φροντίσουμε το ώστε οι μεταφορές και συμφωνώ. Αύριο έχουμε την COP24 και δεν είναι μεταφορές εκεί. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και οικολόγος, είμαι υπέρ ενός φόρου για τη βενζίνη. Δεν ξέρω γιατί δεν ε, ακολουθείτε αυτό. Αλλά τελικά τι κάνουμε, ούτως ώστε αύριο όσοι έχουν πρόσβαση στο αεροπλάνο να πούνε δεν θα πληρώνω πια 20 ευρώ για να πάω από το Παρίσι στη Ρώμη. Ε, μα αυτό είναι. Θα δεχτώ να αναλάβω και το κόστος του οριπένων πληρώνει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, για την Εύα, συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, δημόσιες συγκοινωνίες ούτως ώστε αύριο να έχουμε λιγότερα οχήματα στις πόλεις. Γιατί οι περισσότερες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο στην πόλη γίνονται για αποστάσεις κάτω από 3 χιλιόμετρα. Και, κλείνοντας, ένα πολύ απλό ερώτημα για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε πρώτα τους πειραματισμούς για να αλλάξουμε νοοτροπία και να μοιραζόμαστε πλέον το αυτοκίνητο. Allez, vous allez nous répondre. On commence par qui Ποιο θα απαντήσει πρώτο, ο Φιλίπ. Allez, Philippe, on répond. Ähm, ich kann gerne anfangen. Ähm, Πολύ ευχαρίστω ε, να ξεκινήσω εγώ λόγω του ότι οι περισσότερες ερωτήσεις ετέθησαν στα γερμανικά, θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Και ξεκινάω ε, με το πιο εύκολο και ευχάριστο σχόλιο από τον κύριο Κράμαρ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας για τη δική μου την ιδέα των smart bikes, των εφιών ποδηλάτων. Ε, και εγώ όμως τώρα να σας ρωτήσω, τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε αυτά τα ηλεκτρικά, τα εφή ποδήλατα να στηριχθούν και να προαχθούν. Κάνετε εσείς κάτι. Το ένα είναι αυτό που θέλω να πω. Να συνεχίσω ή θα περιμένω την απάντηση από τον κύριο Κράμερ. Ωραία, να συνεχίσω. Όσον αφορά άλλα ερωτήματα που ετέθησαν, ετέθη το EU ETS, ε, ελέγχθη ότι ορισμένοι άνθρωποι ε, χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για να μετακινηθούν και γιατί να πρέπει να φορολογηθούν ε, αυτοί οι άνθρωποι. Σε τελική ανάλυση το να υπάρχει μία τιμή, ανεξάρτητα με το ποιος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, αυτό δεν είναι σωστό. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να διευκρινίζεται ε, γιατί ε, πρέπει κανείς ε, να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό, αυτό αφορά όλους και εάν είναι ένας ε, ελοχρωματιστής, ε, παραδείγματος που πρέπει να κάνει τη δουλειά του, είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσει και αυτός εναλλακτικέ λύσεις, οι οποίες θα εκπέμπουν λιγότερο διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Από την ε, Καρίν έγινε η παρατήρηση πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα model shift, ε, το να πάμε στο Κατοβίτς, εκεί ε, κοστίζει πολύ λιγότερο. Οι άνθρωποι λένε ότι θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε στην περίπτωση αυτή το τρένο. Εγώ δεν λέω ότι το EU e είναι το μόνο μέτρο, αλλά πιστεύω ότι οι τιμές του EU ETS θα αυξηθούν πάρα πολύ αν συμπεριληφθούν και οι μεταφορές, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ε, στον ε, τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, άρα δηλαδή η διαφορά στις τιμές θα ήταν πολύ ψηλότερες αν επρόκειτο όλα αυτά να ισχύουν για το σύνολο του τομέα των μεταφορών. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποια ερώτηση. Ευχαριστούμε τον Φιλίπ. Η Εύα τώρα έχει το λόγο. Και εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ακόμα φοιτήτρια, δεν είμαι ακόμα εμπειρογνώμων. Έχω διαβάσει μερικά πράγματα και για να τοποθετηθώ στο θέμα του κόστους ε, ε, διάβασα ότι αν υπάρχουν δωρεάν μεταφορές, σε ποιος θα το πληρώσει. Από ό,τι διάβασα, αυτό εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένες ευρωπαϊκές ε, πόλεις και τουλάχιστον στο Ταλίν χρησιμοποιούνται κάποιοι πόροι από τα έσοδα του φόρου εισοδήματος. Υπάρχουν πόλεις που έχουν περισσότερους κατοίκους, αλλά εγώ θεωρώ ότι όλες οι πόλεις θα πρέπει ε, να εφαρμόζουν το μέτρο δωρεάν ε, δημόσιες ε, μεταφορές. Άρα δηλαδή εδώ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίζεται αυτή, αυτό, αυτό το μέτρο δωρεάν μεταφορές. Πάντως, ε, κατά την άποψή μου, σε τελική ανάλυση ε, δεν είναι και τόσο σημαντικό το ε, κατά πόσον πολλούνται εισιτήρια ή όχι, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσανατολιστούμε σε πόλεις όπου οι μεταφορές είναι ήδη δωρεάν. Αυτή την εμπειρία την έχουμε. Υπάρχουν πόλεις που χρησιμοποιούνται ως πειράματα και θεωρώ ότι ο παράγοντας του κόστους, αυτόν τον παράγοντα μπορούμε να τον ξεπεράσουμε και γι' αυτό θεωρώ ότι όλα αυτά είναι εφικτά. Και για να αναφερθώ σε αυτά που είπατε εσείς, δηλαδή το κόστος ε, να προσαρμόζεται στο εισόδημα του ενδιαφερόμενου. Εγώ προσωπικά έχω κάνει την εμπειρία ότι όσοι κερδίζουν αρκετά χρήματα ή να το πω αλλιώ, αν μειωθεί το κόστος για ανθρώπους με χαμηλότερο εισόδημα, να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται ε, με το μετρό, να έχουμε δηλαδή λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, τότε και οι άνθρωποι ε, που μπορούν να το πληρώσουν θα μετακινούνται περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι οι μεταφορές στο σύνολό τους πρέπει να είναι δωρεάν γιατί με τον τρόπο αυτό ε, θα υπάρχει το κίνητρο να χρησιμοποιεί κανείς τις δημόσιες μεταφορές όχι μόνο γιατί δεν έχει αυτοκίνητο αλλά γιατί θα είναι και πιο προσιτό. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο. Βεβαίως ε, ε είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνατε, το να το συγκρίνετε με τη δωρεάν διατροφή, αλλά είναι δύο πράγματα που ε, δεν συγκρίνονται. Και εγώ δεν θέλω να κάνω τη σύγκριση, γιατί ε, για να το κάνω αυτό δεν θα είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου. Σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησης και τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι της συζήτησης ε, που αφορά τον τουρισμό και χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο θα δώσω το λόγο στην Πελουμή Φανταρέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ιδέα μου που αφορά την προώθηση της ιδέας του πολιτιστικού τουρισμού και της βιωσιμότητας. Η ε, βιωσιμότητα εδώ δεν αναφέρεται μόνο στην ε, συντήρηση αλλά και στην ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό και ζητούμε e e, ευφυή και καθολική διακυβέρνηση. Έχουμε έτσι ε, ιδιωτικό δημόσιο τομέα και τους νέους ε, βεβαίως που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα θα πρέπει να γίνονται ε, κοινέ συνεδριάσεις ώστε να κατανοήσουν ε, όλοι τις ανάγκες των μεν και των δε αλλά και να υπάρχει και αυτή η έννοια του ανήκειν. Θα μπορούσε έτσι να φτιαχτεί ένα ειδικό, ένα κόμβος για να μπορούν να συναντιόνται όλοι οι φορείς αυτοί και που θα προσφέρονται ευκαιρίες ε, για να αναπτύσσονται τέτοια μοντέλα, να ε, μεταφέρονται οι ιδέες. Ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμος για να αναπτυχθούν τέτοιες, τέτοιου είδους καινοτόμες συνεργασίες, αλλά και για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλίων αυτών. Γι' αυτό και προτείνω τις εξή δράσεις για να συμβάλλουμε σε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους κατοίκους, τους επισκέπτες και την τοπική κληρονομιά καινοτομία, δηλαδή πρόθεση της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς ε, γεννώντας ε, την υπερηφάνεια για την κληρονομιά αυτή. Δεύτερον, η συμμετοχή στις, στα μαθήματα τέχνης ή ιστορίας με στόχο να χρησιμοποιηθούν οι νέοι ως πρεσβευτές για τους χώρους προστατευόμενους από την UNESCO. Να αναπτύξουν δηλαδή έτσι και υπεύθυνη συμπεριφορά τόσο ως κάτοικοι μιας τέτοιας περιοχής όσο και ως τουρίστες. Τώρα, ε, κοινωνικά δίκτυα. Πολύ ισχυρά, ε, εκεί όπου συναντιόνται όλοι και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μια συμμετοχική διαδικασία για μια κοινή αντίληψη περί κουλτούρας, πολιτισμού, για να ε, αυξηθεί η συνειδητοποίηση όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό. Είναι προορισμός η πολιτιστική κληρονομιά και θα πρέπει ως τέτοιο να εκλειφθεί. Ε, και πιστεύω πως αυτό θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μια αίσθηση του ανήκειν του χώρου που ζει κανείς. Ευχαριστώ πολύ, Πελούμη. Και τώρα το λόγο θα πάρει η Εύα που θα μας μιλήσει για μια άλλη ιδέα που αφορά όμως πάλι τον τουρισμό. Πρόκειται για τις ε, μεταφορές ε, και τον τουρισμό ε, πρόκειται για την επέκταση των ε, μεταφορών με μεταξύ μέτρα. Η τα εισιτήρια να κατέβουν προς το μηδέν και επίσης να υπάρχει διασυνορική συνεργασία διαφόρων μέσων μεταφοράς. Εγώ προσωπικά με την οικογένειά μου ε, ζήσα σε ένα χωριό 300 κατοίκων προς τα γαλλικά σύνορα. Ε, το να μετακινείται κανείς με δημόσια μέσα σε αυτή την περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά τα δημόσια μέσα σε τέτοιες περιοχές μπορούν βεβαίως και να βελτιωθούν και δεν υπάρχει και άμεση σύνδεση με την γειτονική χώρα. Εμείς ε, με την ε, συμφωνία ε, Schengen προχωρήσαμε πάρα πολύ. Έχουμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς, όμως όχι μόνο ανάμεσα σε πόλεις, αλλά και πέρα από τα σύνορα. Αυτό είναι κάτι που θα αναβάθμιζε τις αγροτικές περιοχές, θα οδηγούσε σε πολιτιστική αναβάθμιση και για να παραμείνω στο δικό μου το παράδειγμα, μία γραμμή που συνδέει ένα γαλλικό με ένα γερμανικό χωριό, κατά την άποψή μου θα αποτελούσε μια σημαντική αλλαγή, όπως επίσης και η συνεργασία των ΤΕΖΕΒΕ με την Deutsche Bahn. Αυτό ε, θα μπορούσε ε, να βελτιώσει περαιτέρω την κατάσταση και η σύνδεση επίσης με ε, περιφερειακούς σιδηρόδρομους. Αυτό ε, θα βοηθούσε όχι μόνο εμένα που δεν φταίω σε τίποτα όπως και πολλοί άλλοι, αλλά θα βοηθούσε και άλλους που πρέπει να αποφασίσουν. Οι ε, τιμές ε, θα πρέπει να φτάσουν σταδιακά προς το μηδέν, να εκμεταλλευτούμε προσφορές τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους. Θεωρώ ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να προκύψουν από νέα ταμεία αλλά και από ε, καινούργια που θα συσταθούν. Στο μέλλον να υπάρξει μια αναδιανομή των κονδυλίων και πέρα από αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και αναδιανομή των ε, κοινοτικών κονδυλίων γιατί και αυτά είναι περιορισμένα και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί που χρήζουν επενδύσεων. Eva, une autre idée, Pelumi, c'est à toi. Thank you. The idea today is Η δεύτερη ιδέα σήμερα είναι η δημιουργία ευαισθητοποίηση για τον οικολογικό τουρισμό εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, ποτέ δεν είχα σκεφτεί τον αντίκτυπο που προκαλώ όταν ε, ταξιδεύω. Όμως επισκέφθηκα τη Μαγιόρκα. Και μετά την είχα και μια εμπειρία στη Σλοβενία με τον οικολογικό τουρισμό το 2016. Πολλοί όμως δεν σκεφτόμαστε τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια μας και με τον οικολογικό τουρισμό. Πρέπει στο μέλλον λοιπόν να αυξήσουμε τον οικολογικό τουρισμό για να έχουμε και πιο βιώσιμο τουρισμό. Προτείνω λοιπόν τι εξή ενέργειες. Να δημιουργήσουμε εκστρατείε ευαισθητοποίηση για να αναδείξουμε την ευθύνη που έχουμε όλοι ως Ευρωπαίοι πολίτες στα ταξίδια μας και να προαγάγουμε δραστηριότητες και πρακτικές όπως ο εκλογικό τουρισμός. Να εξετάσουμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στα ταξίδια μας και να ενθαρρύνουμε ε, την ε, βιώσιμη συμπεριφορά και νοοτροπία. Να δώσουμε στήριξη για την έρευνα με χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα προκειμένου τα κρατη να εντοπίζουν και να μετρούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της λήψη αποφάσεων και έτσι να οδηγηθούμε στη βιωσιμότητα. Τέλος, είναι ρεαλιστική ιδέα του οικολογικού τουρισμού γιατί προάχει και την ευημερία του τοπικού πληθυσμού, ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ήπεθρο αλλά και εκτός και να εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες σε κάθε μορφή τουρισμού, το οποίο θα οδηγήσει και στην διατήρηση του περιβάλλοντος. Όμως για να είναι επιτυχής αυτή η διαδικασία πρέπει να έχουμε ε, πολλά ενδιαφέροντα μέρη, όχι μόνο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και ε, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον τοπικό πληθυσμό. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος ε, στους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Βαντεκάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προσωπικά, εμένα μου αρέσουν πιο πολύ αυτές οι ιδέες ε, από τις ιδέες του πρώτου γύρου. Συμφωνώ με την ε, Πελούμε, αν προφέρω στα το όνομά της, ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ε, έμφαση στον βιώσιμο τουρισμό. Βέβαια και εδώ υπάρχει το δύσκολο ερώτημα. Έχουμε να κάνουμε με την επικουρικότητα εδώ και βέβαια θέλουμε ε, η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να ε, προωθήσει τον ε, βιώσιμο τουρισμό. Δεν ξέρω, ίσως το κατάλαβα καλά, αλλά εδώ ποιος θα μπορούσε να ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον. Τότε, παλιά που ήμουν και εγώ νέος, πολλά με ενδιέφεραν, πάντως σίγουρα όχι ο βιώσιμο τουρισμό. Εμείς τότε θέλαμε να πάμε στα μπαρ, στι δισκοτέκ, στη Βαρκελόνη λοιπά. Επομένως όλα αυτά αφορούν την νεολαία ή άλλους ε, μεγαλύτερης ηλικίας όπως εγώ. Ναι, Άντορ, μην νομίζεις. Έτσι είναι. Και αυτούς τους απεχθάνομαι, λέει μετά ο κύριος Βαντεκάμπ, δεν ξέρουμε ποιον εννοεί. Τώρα, για την Ήπεθρο είναι σημαντικό πρόβλημα γιατί οι συγκοινωνίες και οι ε, εταιρείε λεωφορείων ε, λειτουργούν με βάση το οικονομικό κέρδος και χρειάζονται επιβάτες γι' αυτό. Εμείς έχουμε ε, κάποιες δομές εθελοντών που έχουν ένα μικρό πούλμαν και το οδηγούν εθελοντές αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο δικό σου ε, πλάνο ή πρέπει να ανοίξουμε κατευθείαν τον κρατικό κορβανά που ξέρεις ότι δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Μετά για τον ε, οικολογικό τουρισμό, νομίζω ότι συνάδει μετά όσο κάνουμε εδώ και η Κλάντια Ταρπαντέλ και η Μοντέρο ε, συνεχώς προσπαθούν να προβάλλουν αυτή την πτυχή του ευρωπαϊκού τουρισμού και το βλέπω αυτό πράγματι ως ευρωπαϊκό καθήκον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες. Ήθελα μόνο να σας πω από έναν οργανισμό τον οποίο, του οποίου προαδρεύω αυτή τη στιγμή που είναι ο Διεθνής Οργανισμός Κοινωνικού και Υπεύθυνου ε, Τουρισμού δηλαδή και βιώσιμου τουρισμού να πω κατά πρώτον στην ε, Δεσποινίδα Φανταρέ να τη ότι στην Ισπανία και το λέω γιατί επειδή είναι νέα εντάξει υπήρχε μεγάλη ε, παράδοση ε, όσον αφορά τους νέους ε, που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική κατάσταση τους δινόταν η ευκαιρία να μάθουν διάφορες τέχνες για τη συντήρηση του οικολογικού και πολιτιστικού ε, της πολιτιστικής χειρονομιάς της ε, πόλης τους. Ε, υπήρχαν οι κύκλοι τέτοιοι κατάρτισης, τύση, χιλιάδες νέοι τότε ε, εκπαιδεύτηκαν ε, και επιμορφώθηκαν και έτσι έγιναν οι πρωταγωνιστές, οι πρωταγωνιστές της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς και της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό που λείπει είναι τα χρήματα. Το πρόβλημα του τουρισμού στην Ευρώπη είναι ότι οι tour operators πιστεύουν ότι η αγορά τα λύνει όλα και άρα λίγα χρήματα δίνονται για τον τουρισμό. Θα πρέπει να δοθούν χρήματα για την εθνική ανάπτυξη την ανάπτυξη της υπαίθρου και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η, προσδοκία, η, δική σας ε ε, ε, ε, πρόταση θα ήταν πολύ καλή. Εγώ προέρχομαι από μια ζώνη της Υπέθρου και από μια συγκεκριμένη πόλη ε, η οποία κάνει μεγάλες προσπάθειες, μιλάμε για τα δημόσια, μέσα μεταφοράς, ε, συχνά είναι τα ε, αυτοκίνητα του σχολείου, τα σχολικά αυτοκίνητα που μπορεί να ρηπαίνουν. Από ό,τι κατάλαβα στη Γερμανία δεν είναι έτσι, αλλά σε εμά είναι κάπως μονοπωλιακή κατάσταση και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και θα προσπαθούμε όντως να το ε, βελτιώσουμε. Για τον τουρισμό να πούμε ότι υπάρχει ε, κάποιες φορές υπερβολικά πολύ τουρισμός, το είδαμε στη Βαρσικελόνη, το είδαμε στο Παρίσι. Το θέμα είναι να κατανεμηθεί η τουριστική ζήτηση ώστε να υπάρξει περισσότερη βιωσιμότητα. Ποιο άλλο θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριο Δημασμέκερ, όχι. Ωραία. Η κυρία Μάισνερ ήθελε, όχι. κύριο Κράμερ, τότε εσεί θα πάρετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ πολύ ο τουρισμός μπορεί να καταστρέψει τον τουρισμό. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να είναι βιώσιμος. Αλλιώς ο τουρισμός ο ίδιος θα καταστρέψει τον τουρισμό. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε λίγα χρήματα. Έχουμε πολλά χρήματα μόνο που τα δαπανάμε λάθος. Παράδειγμα, στη Στουτγάρδη δαπανώνται 10 εκατομμύρια για να μειωθεί το δυναμικό ενός συντροδρομικού σταθμού μέχρι και το ίμιση. Τρελό, αλλά είναι αλήθεια. Εδώ και 30 χρόνια δαπανάμε δισεκατομμύρια για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου και πέρα από τα σύνορα και αυτό που έχει προκύψει στη πραγματικότητα είναι ένα μπάλωμα ε, γιατί με αυτά τα χρήματα που δαπανώνται θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε όλα τα διοσυνοριακά προγράμματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην περίπτωση αυτή ε, η Ευρώπη θα προχωρήσει προχωρούσε. Ε, και αυτό θα ήταν και οικολογικά πολύ σωστό. Όσον αφορά τον τουρισμό, ε, πρέπει να είναι βιώσιμος ο τουρισμός, το στηρίζω και εδώ έχουμε προχωρήσει στην Ευρώπη πολύ περισσότερο από ό,τι τα κράτη-μέλη. Πάμε το χάνει στην Ευρώπη, δαπανάμε πολλά χρήματα για τις υποδομές, ε, για ποδηλατόδρομους, βεβαίως και αυτό είναι βιώσιμο. Στην Γερμανία η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τέτοιους ποδηλατόδρομους μεγάλων αποστάσεων. Εμείς στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε προχωρήσει πιο πολύ και έχουμε επίσης επιτύχει τα χρήματα να δαπανώνται και αποφασίσαμε επίσης ε, σε, όλα τα τρένα να μπορεί κανείς να παίρνει και το ποδήλατό του. Αυτός ο συνδυασμός του σιδηροδρόμου και των ποδηλάτων είναι πάρα πολύ καλός και το έχουμε επιτύχει στην Ευρώπη. Ε, τώρα ε, τα κράτη-μέλη θέλουν και αυτά να στηρίξουν τέτοια σχέδια. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό γιατί ένα θετικό παράδειγμα είναι παραδείγματος χάρη ο σιδηρο... μάλλον το τραμ ε, από το Στρασβούργο προς το Κέλ. Οι Γάλλοι αρνιόντουσαν, άλλαξε η κυβέρνηση στη Βάδη τώρα υπάρχει τραμ από το Στρασβούργο στο Κέλ και όπου ε, αντικαθιστά το τραμ ε, τα λεωφορεία αυξάνεται ο αριθμός των επιβατών και αυτό έγινε όχι μόνο στο Στρασβούργο αλλά και στο Ζαρμπρούκεν. Ναι στον τουρισμό αλλά πρέπει να είναι βιώσιμος γιατί αλλιώς θα καταστρέψει τον ίδιο τον τουρισμό ε, και τη ζωή πάνω σε αυτό το πλανήτη και δεν το θέλουμε γιατί θέλουμε και τα παιδιά μας να συνεχίσουν να ζουν καλά σε αυτόν τον πλανήτη. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Άλλο θέλει το λόγο. 30 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Κάτι που άκουσα σε σχέση με την δωρεά, τις δωρεάν ε, δημόσιες μεταφορές της πόλης όταν μιλάμε για δωρεάν, κάποιος το πληρώνει. Το πληρώνει η κοινότητα, οι φόροι μας. Το θέμα είναι όταν έχουμε κοινότητες, κυβερνήσεις που δεν θέλουν να πληρώσουν για τα κοινωνικά, τις κοινωνικές παραχές, δηλαδή για τον οικοτουρισμό της ε, κατοικήσιμες πόλης. Ε, δεν είναι το, τα κοινωνικά ζητήματα γενικότερα, δεν το πληρώνουν οι νέοι, αλλά το πληρώνει όλη η κοινωνία. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως από τους φόρους όλων των πολιτών στην κάθε χώρα. Πρέπει λοιπόν να ανακατανεμηθεί ο πλούτος κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ για τις προτάσεις σας για τον οικοτουρισμό που είναι μια από τις προτεραιότητες της της ε, Επιτροπής μας ε, να σας πω ότι έχουμε μια task force στον τουρισμό αν γίνει δεν μπορούμε να τον κάνουμε με αυτοκίνητο όταν θέλουμε να ανακαλύψουμε μια πόλη είναι είτε με τα πόδια είτε με το ποδήλατο αλλά εσείς πώς ε, φαντάζεστε τον μελλοντικό τουρισμό μόνο φέτος η Ευρώπη δέχτηκε, υποδέχτηκε περισσότερους από τους κατοίκους της 600 εκατομμύρια τουρίστες σε ένα χρόνο εμείς είμαστε 500 τουρίστες. Αύριο μεθαύριο θα είναι ακόμη περισσότεροι. Τι κάνουμε. Το έχουμε σκεφτεί αυτό για να διατηρήσουμε όντως τον οικοτουρισμό. Για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο και την Ευρώπη. Είναι ζήτημα και αυτό. Και οι περιοχές της Υπέθρου είναι σημαντικές. Έχουμε την κουλτούρα όμως και την ιστορία των απολύων. Σας δίνω σύντομα το λόγο για να απαντήσετε στους διάφορους βουλευτές. Η Θα σας απαντήσω στα ισπανικά, αφού μου μιλήσατε στα ισπανικά. Μου αρέσει που θέλετε να δώσετε πρωταγωνιστικό ρόλο στους νέους και είναι αλήθεια, είμαστε εδώ, θέλουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στο θέμα του ε, βιώσιμου ε, τουρισμού. Ναι, Τι μου είπατε πριν, είπατε για σχολεία, για σχολεία και για μαθητείες. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους να μάθουν τι είναι η πολιτιστική κληρονομιά, να ταυτιστεί με αυτήν και να κατανοήσει είναι και πολύ σημαντικά τα κοινωνικά δίκτυα. Τα πάντα γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι δημιουργείται περισσότερη συνειδητοποίηση και γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει και μας ε, επιτρέπει και εμάς τους νέους, ε, γιατί είναι πιο εύκολο να ασχοληθούμε και να καταλάβουμε ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι πολύ σημαντικός και αφορά την ε, πολιτιστική μας κληρονομιά και πρέπει αυτή να την προσέξουμε πάρα πολύ. Και τώρα θα απαντήσω στον κύριο Κράμπ, εσείς ε, ρωτήσατε για το βιώσιμο τουρισμό, ποιο είναι δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος ε, της Ένωσης σε αυτό. Ε, είναι σίγουρα αλήθεια, είναι κάτι που οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να το δουλέψουν γιατί εξαρτάται άμεσα από εκείνες, αλλά θα πρέπει προς τους νέους να μιλήσουμε και να φτιάξουμε ε, έτσι οι νέοι να αποκτήσουν γνώση ε, και να ενημερωθούν. Εάν υπάρχει αυτή η ιδέα και προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πολύ καλύτερο πιστεύω. Για τα χρήματα ρωτήσατε και δώσατε το παράδειγμα του Φράιμποργκ που έχει πολλά χρήματα αλλά δεν τα χρειάζεται. Θα έπρεπε ίσως να σκεφτούμε ε, πού πάνε τα χρήματα, ποιες πόλεις, άλλοι... Ε, ε Ποιε άλλε πόλει θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα και γι' αυτό και ανέφερα την ιδέα των ερευνητών. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε περισσότερο σε ερευνητέ και δεδομένα για να γνωρίζουμε πού πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα και πού πραγματικά θα χρησιμεύσουν ώστε να μην χάνονται κονδύλια. Ευχαριστώ. Η Εύα. Ja, wieder auf Deutsch. Ähm, Θα μιλήσω γερμανικά και πάλι. Καταρχήν, όσον αφορά τη χρηματοδότηση και το θέμα της ε, ε, απόδοσης, ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και ίσως και να είναι το σημαντικότερο αντεπιχείρημα. Όπως σας είπα, εγώ έρχομαι από αγροτική περιοχή και έχω κάνει ακριβώς αυτή την εμπειρία, ότι ακόμα και αν υπάρχουν ε, λεωφορεία και σε εμά το δικό μας το χωριό υπάρχουν λεωφορεία, αυτά είναι σχεδόν πάντα άδεια. Γι' αυτό λοιπόν πρότεινα δύο πράγματα. Πρώτον, να μειωθούν οι τιμές των εισιτηρίων και δεύτερον, να βελτιωθούν οι μεταφορές στις αγροτικές περιοχές. Στη δική μου την περιοχή, αν έχει κάποιος αυτοκίνητο που δεν έχουν όλοι, αποφασίζει να το χρησιμοποιήσει υπέρ του αυτοκινήτου. Ε, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όσον αφορά το κόστος, ε, ξέρετε, στο λεωφορείο πάνε όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και είναι κάτω τη ηλικία των 18 ετών. Αλλιώ δεν αξίζει να χρησιμοποιεί κανείς το λεωφορείο. Άρα δηλαδή πρέπει ε, να μειωθούν οι τιμές ε, των λεωφορείων γιατί στη δική μου την περιοχή είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Αυτό οφείλεται ε, στις, στους δήμους, στις κοινότητες. Κάτι πρέπει να γίνει, να μην γίνουν βέβαια όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχω καταλάβει πολύ καλά. άκουσα με μεγάλη μου χαρά ότι ε, εντωμεταξύ υπάρχουν ε, κάποιες εξελίξεις. Ε, παραδείγματος χάρη ότι μπορεί κανείς να παίρνει αυτοκίνητό του στο τρένο. Μεγάλο χειροκρότημα για τους νέους μας λοιπόν. Merci pour cet échange. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ όποτε θέλετε. Αλλά όχι την ώρα στο Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και είμαστε ευτυχείς που η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τους νέους μονιμοποιείται και γίνεται κάθε χρόνο. Είμαστε μεγάλοι υποστηριχτές. Ευχαριστούμε και στο Πανεδίνα. Allez, nous continuons nos débats et nous allons dire... Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα τι συζητήσει μα Θα περάσουμε απευθεία στο επόμενο θέμα, η έκθεση για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση του κυρίου Keith Taylor. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ενεργό συμμετοχή του στην κατάρτιση αυτή της ε, γνωμοδότησης για τον κανονισμό 1 του 2005. Παρότι υπάρχει μια διαφορά απόψεων, ε, όπως καταδεικνύεται και από τις 90 τροπολογίες που έχω λάβει. Πολύ λυπάμαι που έχει περάσει μια δεκαετία από την ε, υιοθέτηση και θέση ισχύ του κανονισμού και έχουμε ακόμα ε, τις ίδιες παραβιάσεις που καταγράφονται ξανά και ξανά. Οι περισσότεροι συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες για τη βελτίωση της ευημερίας των ζώων. Ε, και εδώ πρέπει να βρούμε συμβαστικές ε, λύσεις για την καλύτερη υλοποίηση, ισχυρότερους μηχανισμούς ε, εφαρμογής του νόμου και ισχυρότερες κυρώσεις. Εμείς εδώ σε Επιτροπή Μεταφορών εξετάζουμε και συγκεκριμένες τεχνικές βελτιώσεις για τον εξοπλισμό θαλάσσιων και οδικών μεταφορών. Οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει μείωση του χρόνου μεταφοράς των ζώων και αύξηση ε, των ε, ελέγχων πριν από την φόρτωση. Άλλοι λένε ότι ο κανονισμός ε, δεν γίνεται σεβαστός εξαιτίας των εξαγωγών σε, κατά τη διάρκεια εξαγωγών σε τρίτες χώρες παρά τη δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκές διατάξεις να γίνονται σεβαστές μέχρι τα ζώα να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, ακόμα και αν αυτό είναι σε τρίτη χώρα. Μέχρι τώρα λοιπόν, ακόμα προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Κανονικά θα ψηφίζαμε αύριο, αλλά κάποιες πολιτικές ομάδες ε, επανήλθαν και είπαν ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα ψηφίσουμε λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, στις 3 Δεκεμβρίου. Πριν από αυτό θα γίνει την επόμενη Δευτέρα και μία συνάντηση των Σκιωδών στις 26 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Θα θυμάστε ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη υιοθετήσει ψήφισμα για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους το 2012. Δεν νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να επαναλάβουμε αυτή την έκκληση στο κείμενό μας ούτε εννοείται να έχουμε ένα ακόμα πιο αποδυναμωμένο κείμενο. Ο έξω κόσμος θέλει να δει από τα αποτελέσματα, γιατί πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες ε, είχαν υπογράψει μία εκτρατεία για την απαγόρευση όλων των μεταφορών ζώων για πάνω από 8 ώρες. Εδώ λοιπόν θέλουμε να δούμε πραγματική ανάληψη δράσης. Και έχει έρθει η ώρα λοιπόν για φιλόδοξα σχέδια. Γιατί λοιπόν να αρκεστούμε στο status quo, το οποίο δεν λειτουργεί καλά και έχουμε ακόμα τέτοια φαινόμενα που τόσα πολλά ζώα ε, υφίστανται ε, απαράδεκτες ε, συνθήκες και υποφέρουν. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες ε, και ελπίζω να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί με τους συναδέλφους. Θα στείλουμε λοιπόν τις προσκλήσεις ε, στους συναδέλφους ε, σήμερα. Προς το παρόν λοιπόν απλώς περιμένω να ακούσω τις ε, παρατηρήσεις σας. Αν θέλετε να συμπεριλάβουμε κάτι στις προτάσεις συμβασμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους Κιώδης και στα υπόλοιπα μέλη να καλωσορίσουμε τον ε, Δήμαρχο του Λιβέρνου. Πού βρίσκεστε? Σηκωθείτε παρακαλώ. Ο κύριος Φίλιππο Νογκαράν. Καλώς ήρθατε. Από την Ιταλία λοιπόν. Συνεχίζουμε. Κύριε Ντελή. Έχετε το λόγο ξανά από της κυρίας Ντεμόντε. Της κυρίας Μοντέρο μάλλον. Παραλίγο διπλωματικό επεισόδιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η κυρία Μοντέιρο μου ζήτησε ε, να σας μεταβιβάσω την τοποθέτησή της, γιατί δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα εν γέρος. Πρώτα απ' όλα, So far, uh, before making some comments on the compromise amendments, I would like to underline... Πριν σχολιάσω τις συμβαστικές τροπολογίες, ε, να επισημάνω ε, τη θέση του ΕΛΚ. Θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη εφαρμογής του νόμου από τα κράτη-μέλη ε, και έλλειψη ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία περιφέρεια του κόσμου δεν έχει τόσο ε, αυστηρή και ολοκληρωμένη νομοθεσία για την επιμερία των όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέσα επιβολής του νόμου σε όλη την αλυσίδα για να ε, εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι πριν από την ανάληψη δράση θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Κομισιό να παρουσιάσει τις μελέτες σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας. Όμως, οποιαδήποτε απαγόρευση στα μακράς διάρκειας ε, ταξίδια θα πρέπει να ε, ακολουθείται και από ε, μελέτη αντικτύπου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις επιμέρους πλατφόρμες ε, που ασχολούνται με την ευημερία των ζώων όλους μας ενδιαφέρει φυσικά η ευημερία των ζώων, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, όλους τους παράγοντες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, με μεγαλύτερη αυστηρότητα να ελέγχουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται και να διεξάγονται και αναλογικέ επιθεωρήσει, όπω αναφέρεται και στην νομοθεσία. Απαιτείται και καλύτερη συνεργασία μεταξύ ε, ευρωπαϊκών χωρών και τρίτων χωρών. Και πρέπει ε, να παρέχεται και αρρωγή για την ε, παρακολούθηση και τη συμμόρφωση. Κλείνοντας, αφενός χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση, κατάρτιση, διάδοση βέλτιση των πρακτικών. Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να κινηθεί κατά των κρατών μελών που συστηματικά ε, δεν τηρούν τον κανονισμό. Ελπίζω αυτή η παρέμβαση ε, να συμβάλλει και στην κατάρτιση συμβαστικών τροπολογιών για να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο. Ευχαριστώ. Monsieur Ευχαριστώ κύριος Ζίνκε. Ε, ε, Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένε παρατηρήσει. Εξ ονόματο της πολιτικής μου ομάδα. Εμείς δεν εστιάζουμε την προσοχή μας την κατάρτιση μιας νέας νομοθετικής πράξης. Θέλουμε απλώς ε, μια αξιολόγηση του κανονισμού που υπάρχει εδώ και μερικά χρόνια. Υιοθετήθηκε το 2005. Γι' αυτό και θα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού μπορεί να είναι θετική. Η απάντηση είναι όχι, δυστυχώς η πολιτική μου ομάδα δεν έχει θετική αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, οι νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να καλύπτουν όλες, όλους τους τρόπους μεταφοράς. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις θαλάσσιες μεταφορές, ε, όπου η έλεγχη είναι σίγουρα πιο πολύπλοκη από ότι στις οδικές μεταφορές. Δεύτερον, τα ζώα θα πρέπει να την χάνουν και της κατάλληλης κτηνιατρικής φροντίδας. Τρίτον, είμαστε πεπισμένοι ότι οι έλεγχοι δεν πρέπει να αφορούν μόνο τις εισαγωγέ και εξαγωγέ στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής επικράτειας. Αντίστοιχη υποχρέωση και ηθική υποχρέωση μάλιστα υπάρχει και για τον έλεγχο των μεταφορών ε, από τις ε, ευρωπαϊκές χώρες και προς τις τρίτες χώρες. Κάποιες φορές κατανοώ από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ότι ε, οι συντάκτες τους έχουν πολύ αγαθές προθέσεις, αλλά δεν είναι ρεαλιστικές. Πώς γίνεται κάθε ε, ζώο που μεταφέρεται μπορεί να έχει ένα τσίπ. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είστε επιφυλακτικοί με αυτές τις ιδέες, γιατί μπορούμε να ε, το φανταστούμε στις αγελάδες ε, και στα άλογα, αλλά στα πουλερικά, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να ισχύσει κάτι τέτοιο. Πρέπει πρώτα λοιπόν να δούμε αν αυτό που προτείνουμε είναι ρεαλιστικό από πρακτική άποψη. Δεν θα ήταν καθόλου καλό να προτείνουμε μη ρεαλιστικέ ε, και μη εφαρμόσιμε νομοθετικές διατάξεις. Εγώ, όπω και η πολιτική μου ομάδα, είμαστε ανοιχτά διακείμενοι προ την εξέβρεση συμβιβασμών είναι πολλές οι συμβαστικέ τροπολογίες. Αν δεν υιοθετηθούν αυτές, τότε θα πρέπει να υιοθετηθεί η γνωμοδότηση με το ζόρι και αυτό δεν θα ήταν θετικό. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση για την εξέβρεση συμβιβασμών. Ευχαριστώ κύριε Ζωτόφσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος του προκαθηγητή Λεγκούτκο. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε εισηγητή για τις ε, συμβαστικές προτάσεις ε, με τις οποίες εν γέννη συμφωνούμε. Οι συμβαστικές αντικατοπτρίζουν την σημερινή κατάσταση της εκτέλεσης ε, του κανονισμού 1 του 2010, 2005 ε, με συγχαρείτε, που σχετίζεται με την προστασία των ζώων στη διάρκεια της μεταφοράς τους. Θα ήθελα να επιμείνω για το γεγονός ότι η, πρόοδη, η πρόοδος στην εφαρμογή του κανονισμού δεν είναι ικανοποιητική. Ε, το πρόβλημα με την ευημερία των ζώων παραμένει λόγω της έλλειψης σε αυστηρή εφαρμογή των κανόνων στα κράτη-μέλη. Η εφαρμογή δεν έχει επαρκώς γίνει σεβαστή. Θα πρέπει λοιπόν να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από την αρχή μέχρι το τέλος των μεταφορών. Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί επιμένουν ότι θα πρέπει να περιοριστεί η διάρκεια των ε, ε, μεταφορών στις 8 ώρες με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνονται οι μεταφορές αυτές. Επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να γίνουν συχνότεροι έλεγχοι ε, και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεριμνήσουμε για την ευημερία των ζώων στη διάρκεια των μεταφορών. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα σύντομα, ώστε η Επιτροπή ε, Γεωργίας να μπορέσει να λάβει υπόψη τη γνώμη μας. Κύριε Μάισνέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Τέιλορ. Έγινε μια ακρόαση για τη μεταφορά των ζώων. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, αλλά μου είπαν ποια ήταν τα εμπόδια στην εφαρμογή του κανονισμού. Εξαιρετικά λίγοι έλεγχοι γίνονται. Υπάρχουν χώρες που προβαίνουν σε ελέγχους, αλλά όχι όλες. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, η νομοθεσία σε σχέση με τα φορτία δεν είναι πάντοτε ε, ε, διαθέσιμη και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εφόσον υπάρξει πρόβλημα υγείας και αν ένας ε, ε, κτηνίατρος πρέπει να παρέμβει. Πρέπει τα ζώα που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις να έχουν νερό και τροφή. Κατά συνέπεια, θα πρέπει τα ζώα να πηγαίνουν στο πιο κοντινό σφαγείο από το μέρος όπου εκτρέφονται. Θα πρέπει να μερεμνήσουμε ώστε τα ζώα που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις να την χάνουν της ε, σωστής περίθαλψης όταν έχουμε σφαγή των ζώων, αυτό δεν είναι προ το όφελο τη κοινωνία. Αυτό βέβαια μοιάζει να είναι φυσιολογικό προ την κοινωνία μα. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία. Είναι πολύ λίγα τα στοιχεία ε, και πολύ λίγα τα συμπεράσματα που μπορεί κανεί ε, να χρησιμοποιήσει. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί κατ' ουσίαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα ε, των νόμων και αν κάτι ε, δεν πάει καλά, θα πρέπει να μεριμνήσει, όχι μόνο να στέλνει επιστολές, αλλά η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται στα κράτη-μέλη και από ό,τι φαίνεται η εφαρμογή γίνεται με διάφορους τρόπους, όχι πάντα όπως το προβλέπει η νομοθεσία και όχι πάντα ε, προς την ευημερία των ζώων και πρέπει αυτό να το βελτιώσουμε. Όπως επίσης ε, και τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα θα πρέπει να είναι σωστά εξοπλισμένα. Η κυρία Γκονζάλες, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή πέρα από τις δικές μας τροπολογίες θα ήθελα να μιλήσω για το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω πως ε, προχωρούν καλά, αλλά αυτό που λείπει είναι να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αναθεωρήσει το σύνολο του κανονισμού για την ευημερία των ζώων ε, στη διάρκεια της μεταφοράς τους, γιατί τελικά όταν εγκρίναμε αυτή την πρωτοβουλία ε, ήταν πριν 14 χρόνια. και μπορεί και να μιλάμε για άλλα δύο χρόνια μέχρι να εγκριθεί ο επόμενος. Πιστεύω πως σήμερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία προς τα ζώα και ε, όσον αφορά τη μεταχείριση που τους επιφυλάσσουμε. Η Κομισιόν προτίθεται να εξυγχρονίσει κάποια πράγματα, όμως πιστεύω πως το καλύτερο θα ήταν μια πλήρης αναθεώρηση. Εν τω μεταξύ χαιρετίζουμε θετικά ε, καταρχάς ε, το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει ε, γιατί οι σημερινές τεχνολογίες είναι αρκετά προηγμένες όσον αφορά την, τον γεωγραφικό εντοπισμό μέσω δορυφόρων για να μπορούν να εντοπίζονται ζώα είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες. Μπορεί κάτι τέτοιο να έχει υψηλό κόστο, αλλά πρέπει να το αξιολογήσουμε για να κάνουμε και οικονομίες κλίμακας, ε, να αναλάβουμε ας πούμε, αυτό ε, για λογαριασμό των ε, μικρών κτηνοτρόφων από πλευρά μα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτό το σύστημα, αλλά πιστεύω πω θα άξιζε τον κόπο. Επίση, ω κυρώσει θα έπρεπε να αποσύρονται οι άδειε στου κτηνοτρόφου που δεν σέβονται αυτέ τι νομοθεσίε, όπω συμβαίνει σε χώρε όπω η Αυστραλία. Να πω επιπλέον ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη με την πρόταση των συναδέλφων να δημοσιευθούν οι μαύρε λίστε ε, που υπάρχουν ήδη για του διάφορου ε, που δεν τηρούν την οδηγία για την ώρα αυτά έχω να σας πω. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, γιατί πρέπει να πάω και σε άλλη μια συνεδρίαση, αλλά θα ακούσω τις απαντήσεις σας και θα τις λάβω υπόψη μου. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Madame εδώ μιλάμε για την ε, εγκληματική αμέλεια απέναντι στα ζώα στη διάρκεια των μεταφορών. Οι περισσότερες ε, τροπολογίες ε, είναι θετικές ε, και τις βλέπει θετικά ο εισηγητής, όπως ας πούμε αυτή για τα κινητά σφαγεία, πράγμα που δεν εξαρτάται από τη δική μας Επιτροπή, αλλά που είναι πολύ σημαντικό γιατί εν μέρη θα έλυναν το πρόβλημα της μεταφοράς των ζώων σε αβάσταχτες συνθήκες. Αλλά οι περισσότερες τροπολογίες κατευθύνονται στη σωστή κατεύθυνση, Ωστόσο, υπάρχουν και δύο βασικά ζητήματα που αφορούν αυτό εδώ το θέμα. Πρώτον, αντίληψη του πολιτισμού μας για το ζώο, και για, για ένα ζωντανό οργανισμό αγνοείται ή παραμελείται η ευημερία του ε, ενός ευαίσθητου όντως. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη φύση της ευρωνίας αγορα η οποία είναι στραμμένη αποκλειστικά προς το κέρδος ε, και που καταλήγει σε όλο ένα και πιο μεγάλες αποστάσεις μεταφορών για τα εμπορεύματα όπως είναι και τα ε, ζώα. Τα ζώα θεωρούνται μόνο σε εμπορεύματα και ε, αυτό εις βάρος οποιοδήποτε ε, περιβαλλοντικού ή κοινωνικού κόστους. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να διατηρηθεί αυτή η εκμετάλλευση των ζώων είναι αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν και τους οδηγούς των φορτηγών. Ευχαριστώ. Τόμας Μίκε. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Δεμές Μάκερ. Και για μένα είναι πολύ σημαντικά τα ζώα βέβαια. Όπως ε, ανέφεραν ε, οι συνάδελφοι και ο κύριος Τέιλορ και άλλοι συνάδελφοι και εγώ με τα λύπης βλέπω την ε, ελλειπή, και διαπιστώνω την ελλειπή εφαρμογή του κανονισμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά ζώων. Είναι πραγματικό σκάνδαλο το να μην μπορούμε να ελέγξουμε ή να μην θέλουμε να ελέγξουμε ε, την εφαρμογή της νομοθεσίας μας, τότε όλη αυτή η πολύ καλή νομοθεσία που έχουμε, τι είναι ε, ένα χαρτί. Είναι ένα θέμα το οποίο επανειλημμένως ε, έχει επισημανθεί στο Animal Welfare Intergroup του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή ήταν και, και στην Επιτροπή μας και συζητητής ε, για αυτό το θέμα. Χαίρομαι που η Επιτροπή μας λοιπόν έχει μια γνωμοδότηση. Υπήρχαν κάποιες τροπολογίες ε, οι οποίες ε, αναφέρθηκαν στην πρώτη συνάντηση των σκιωδών και λυπάμαι που δεν τις υποδέχθηκαν όλοι με τόση θέρμη. Ωστόσο και οι τροπολογίε του κυρίου Τέιλορ και άλλων συναδέλφων είναι να βγούμε προ τη σωστή κατεύθυνση, να περιορίσουμε τον χρόνο μεταφοράς, ε, να το επεκτείνουμε και στι εξαγωγέ εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωση, προ χώρε χώρες ε, και η, η επιβολή και η εφαρμογή τη νομοθεσία είναι βασικά στοιχεία. Ελπίζω η συγκεκριτή μαζί με του κοιότητε να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία για αυτό το σημαντικό φάκελο. Ευχαριστούμε. Κυρία Χουισκόφ. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Εδώ και καιρό το θέμα της μεταφοράς ε, ζώων μας απασχολεί. Έχουμε όλοι δει φρικτές εικόνες Όμω, η συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στο παρελθόν έχουμε δει ότι υπάρχει πολύ σημαντική κακοποίηση ζώων κατά τη διάρκεια τη μεταφορά του Μεταφέρονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπό φρικτέ συνθήκες. Και οι Ευρωπαίοι πολίτε εδώ και πολύ καιρό έχουν ε, δηλώσει τη δυσαρέσκειά του όταν βλέπουν αυτές τις εικόνες στην τηλεόραση, όταν τα ακούν όλα αυτά στο ραδιόφωνο, πραγματικά θορυβούνται. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τις μεταφορές ζώων και Ελπίζω να υπάρξει πλειοψηφία υπέρ αυτής της πρότασης και ελπίζω και οι τροπολογίες μου να λεφθούν υπόψη στις συμβαστικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή συνεργασία. Είναι μια πολύ καλή έκθεση και νομίζω ότι θα επιτύχουμε την πλειοψηφία στην ψηφορία. Οι μεταφορές ζώων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για ζώντα ή σφαγιασμένα ζώα. Παράδειγμα, οι ε, καραβίδες στην Νορβηγία και στην Βόρεια Θάλασσα μεταφέρονται στο Μαρόκο γιατί εκεί οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, τις επεξεργάζονται και μετά τις ε, επαναφέρουν πάλι αυτές τις καραβίδες ε, στο βορρά. Αυτό είναι τρελό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα ζώα, τα οποία μεταφέρονται στα πιο κοντινά σφαγεία. Τη δεκαετία του 40 και του 50 ήταν μικρές οι μεταφορές, οι αποστάσεις, αλλά τα μεγάλα σφαγεία ήταν πιο φτηνά, έκλεισαν τα μικρά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μεταφορές των ζώων. Μεταφέρονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα και αυτό το κρέας επανέρχεται εκεί που κατ' ουσίαν πρώτα προέκυψε. Είναι τρελό γιατί ε, αυτό προκύπτει και διότι οι μεταφορές ε, γίνονται πιο φθηνές. Άρα δηλαδή μην εκπλήσεστε για τα αποτελέσματα, πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Και θα ήθελα να γνωρίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν κάνετε τίποτα εδώ και χρόνια. Εσείς είστε θεματοφύλακες των συνθήκων, παραβιάζονται οι συνθήκες και ένας ε, νόμος που κανείς δεν τον ελέγχει και δεν προβλέπονται κυρώσεις, ξεχάστε το. Πρέπει να ξέρετε, ένας νόμος έχει νόημα μόνο όταν γίνεται σεβαστό στην πράξη και όταν υπάρχουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ευχαριστώ. Στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Ραμίρες Μπέλα. Την Τίτζη Σαντέ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προσήλωση εργάζεται για τη βελτίωση της εφαρμογής ε, της υφιστάμενης νομοθεσίας Υπάρχουν και ενέργειες αυτή τη στιγμή για να αποκομίσουμε μια ευρύτερη εικόνα για τις ε, οδικές μεταφορές και εξαγωγές, αλλά και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Και άλλες δράσεις συνεχίζονται για τις μεταφορές σε υψηλές θερμοκρασίες και εξαγωγές σε τρίτες χώρες και δράσεις για την διαθεσιμότητα των δεδομένων που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε κρίσιμη σημασία τομείς για την ευημερία των ζώων. Θεωρούμε ότι υπάρχει σωστή εφαρμογή του κανονισμού διασφαλίζεται η ευημερία των ζώων και ε, περιμένει με ενδιαφέρον ε, την τελική έκθεση της Επιτροπής σας για να ακούσουμε και με προσοχή τις συστάσεις που θα απευθύνεται προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ ο κύριος Κίστελοχ. Ο κύριος Keith Taylor, μάλλον, είναι η πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίες οι παρεμβάσεις σας. Ε, πραγματικά Πολύ χαίρομαι που φαίνεται να συμφωνούμε σε τέτοιο βαθμό ότι η εφαρμογή είναι ελλειπής. Τώρα λοιπόν το θέμα είναι πώς θα έχουμε την καλύτερη δυνατή βελτίωση της κατάστασης. Πώς θα βρούμε λύσεις που όπως είπαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες νομίζω θα είναι ε, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Απογοητεύομαι λίγο βέβαια από την άλλη που στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Δεν αναγνωρίζουν ότι εκείνοι είναι θεματοφύλακες ε, των συνθήκων. Είναι εύλογο να περιμένει κανεί ε, να ακούσει από την Επιτροπή τι κάνει ακριβώ για την επίλυση του προβλήματο. Δεν φτάνει η συλλογή δεδομένων. Εδώ και 10 χρόνια μπορεί να μαζεύεται δεδομένα. Αν το κάνατε μέχρι τώρα θα είχαμε επαρκή δεδομένα σίγουρα. Δεν θα χρειαζόμασταν άλλα. Θα καταγράψω λοιπόν και θα λάβει υπόψη όλες αυτές τις ε, παρεμβάσεις και αυτή την πρόταση ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απομιστούν ε, εν μέρη το βάρος για τα περιφερειακά ή τα κινητά σφαγεία. Και κάπως θα πρέπει να αξιοποιηθεί εδώ το Ταμείο Συνοχής, κατά τη γνώμη μου. Γιατί νομίζω ότι έτσι θα ε, ήταν μια δίκαιη λύση για όλους. Όμως, πίσω από όλα αυτά κρύβεται το εξή θέμα. Ο ανθρωπισμός μας ε, εξαρτάται και καθορίζεται και από τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα ζώα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να τους φερόμαστε με τέτοιο ε, φρικτό και απάνθρωπο τρόπο όπως κάνουμε σήμερα. Θα εξετάσω λοιπόν ε, τις τροπολογίες, θα ξανασυζητήσουμε με τους κοιόδης την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Donc, le vote Λοιπόν, η αρχική ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για την επόμενη εβδομάδα. Θα αναβληθεί όμω ε, για μεταγενέστερη ημερομηνία. Συνεχίζουμε με την έκθεση της κυρίας Μαρίτα Ούλσκοχ Θερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας». Γεια σας κύριε Σβόμποντα, καλώς ήρθατε. Παρακαλώ, λόγο στην κυρία Συγγετρία. Α, όχι. Πρώτα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Χαουγκάρτ, είστε έτοιμος να μας μιλήσετε για την αλλαγή της ώρας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, Αγαπητοί συγγητροί, αγαπητά μέλη, ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτήν την Επιτροπή για να σας παρουσιάσω σύντομα την πρόταση της Επιτροπής ε, ε, σχετικά με το να μην υπάρχουν πια αυτές οι αλλαγές στην ώρα, στην περί... να αναφερθώ στην περίφημη οδηγία περί θερινής ώρας. Εχθές έγιναν τριμερείς διάλογοι για θέματα που αφορούν στον τομέα της αεροπλοείας και έχουμε πάρα πολλά καλά νέα από αυτά. Επανερχόμεθα στη τέννη ώρα. Ξέρουμε ότι ο κύριος Γιούγκερ στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ένωση έκανε αυτή την πρόταση και αυτό για να δείξει ε, την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε θέματα επικουρικότητας και για να αποδείξει επίσης ότι θα υπάρχουν και υπάρχουν ρυθμίσεις μόνο όταν προκύπτει σαφής προστιθέμενη αξία και για να αποδείξει επίσης ε, στους πολίτες μας ότι πραγματικά ακούμε τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους γιατί στην περίπτωση ε, των, ε, της αλλαγής της ώρας ε, δεν έχει υπάρξει καμία θετική στάση ε, κάθε φορά που οι πολίτες εκλήτησαν να αλλάξουν τα ρολόγια τους, δηλαδή δύο φορές το χρόνο. Να σας πω λοιπόν τι κάναμε. Η δική μου ομιλία ε, περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Πρώτα να σας ε, εξηγήσω ένα μικρό ιστορικό, μετά θα μπω στο περιεχόμενο και τέλος ελπίζω να μπορέσω να σας εξηγήσω πώς ακριβώς βλέπουμε το μέλλον. Όσον αφορά το ιστορικό, όλοι μας γνωρίζουμε το ιστορικό ε, έχουμε δύο φορές το χρόνο, αλλαγή της ώρας. Αυτά ξεκίνησαν από τον στόχο των κρατών μελών, ε, κατά κύριο λόγο, ε, να εξοικονομείται ενέργεια. Αυτά εισήχθησαν από τα κράτη-μέλη έχοντας κατά νου τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Μετά πολλά κράτη εγκατέλειψαν αυτή την ιδέα, αλλά τη δεκαετία του 70 επανήλθαν αυτές οι ρυθμίσεις. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θερινή ώρα εισήχθη για πρώτη φορά το 1980, κατά κύριο λόγο για να διασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση στην κοινή αγορά. Από το 2001 η τερινή ώρα ρυθμίζεται από την 2000 κάθετος 84 κάθετος EC και εκεί αναφέρεται η υποχρέωση όλων των κρατών μελών ε, την τελευταία ημέρα του Μαρτίου να αλλάζουν την ώρα και να επανέρχονται ε, την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου στην χειμερινή ώρα. Ε, γιατί λοιπόν προτείνουμε να καταργηθεί αυτό τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε κυρία Πρόεδρε, ε, πολύ απευθύνθηκαν στην Επιτροπή να το εξετάσει το θέμα και ε, πολλές από τις εκκλήσεις ήρθαν από το Κοινοβούλιο, είδαμε τις επιστολές, υπήρξαν αναφορές που καταχωρίστηκαν, υπήρξαν συζητήσεις στην Ολομέλεια και το Φεβρουάριο μας καλέσατε στο ψήφισμά σας να αξιολογήσουμε την οδηγία και αν κρυφτεί απαραίτητο να κατατεθεί πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας. Και ακριβώς αυτό κάναμε. Δεν ήσασταν μόνοι σας στο να αμφισβητήσετε το ισχύον σύστημα. Είχαμε επίσης και πάρα πολλές ερωτήσεις από πολίτες και ένα αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών. Έτσι λοιπόν αξιολογήσαμε τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Ε, είχαμε και μια πολύ καλή μελέτη επιπτώσεων που έγινε από εσάς τους ίδιους ε, τον Οκτώβρη και σε αυτή την έκθεση αναφέρεται ότι η οι λόγοι πια δεν είναι τόσο αποχρόντες, κυρίως όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Αποδείχθηκε ότι δεν εξοικονομείται πολύ ενέργεια. Και επιπλέον η ε, ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, ε, τα, οι σε μετρητές, ε, με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται περαιτέρω τα ωφέλη. Εξάλλου, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία και εκεί υπάρχει μια ασάφεια, παρότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στην αλλαγή του βιορυθμού του ανθρώπου ίσως είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι πιστεύουμε κατά το παρελθόν. Και για την οδική ασφάλεια, και εκεί δεν υπάρχει σαφήνεια. Πάντως, οι λόγοι γιατί πρέπει να εισαχθούν αυτοί οι κανόνες, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν πια. Και όπου υπάρχουν σαφή στοιχεία είναι η περίπτωση όπου ε, εάν αλλάξουν όλοι μαζί αυτό θα ήταν ζημιογόνο για το εμπόριο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προέκυπταν ε, αναταραχές και το καθεξής. Εμείς λοιπόν καταλήξαμε ε, στο ότι όπως ξέρετε μετά από ε, διαβουλεύσεις ε, και από εκεί προέκυψε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις και πάνω από το 99% ήρθαν από πολίτες. Αυτές είναι οι περισσότερες αντιδράσεις που είχαμε ποτέ σε μια δημόσια διαβούλευση. Το 84% είναι υπέρ του να καταργηθεί αυτή η αλλαγή της ώρας και οι περισσότεροι αναφέρουν ε, το επιχείρημα της υγείας. Μετά άλλοι λένε ότι δεν εξοικονομείται ενέργεια. Παρότι βέβαια δεν απόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίζει, εμείς ε, ρωτηθήκαμε αν τελικά καταργηθεί αυτή η αλλαγή της ώρας ε, τι θέλουν οι πολίτες ε, την θερινή ώρα ή την standard ώρα και το 56% είπαν ε, την μόνιμη θερινή ώρα το 36% την μόνιμη χειμερινή ώρα και 8% είπαν δεν έχουν καμία προτίμηση. Άρα δηλαδή με όλα αυτά τα στοιχεία κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της και τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι τα εξής. Και τώρα μπαίνω στην πεμπτουσία της πρότασής μας. Προτείνουμε να μην αλλάζει πια η ώρα σε όλα τα κράτη-μέλη από την 1η Απριλίου του 2019. Και το 19 θα αλλάξουν όλοι στις 31 Μαρτίου ε, σε θερινή ώρα. Τα κράτη-μέλη όμως που επιθυμούν να επανέλθουν στη χειμερινή ώρα μπορούν να το κάνουν αυτό ε, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Ε, με βάση τους... Συγγνώμη, να τα ξαναπείτε, λέει η Πρόεδρος, γιατί δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, προτείνουμε να μην υπάρχουν αλλαγές στην ώρα σε όλα τα κρατη από την 1η Απριλίου του 2019 και μετά θα γίνει η αλλαγή από όλους στις 31 Μαρτίου. Βέβαια, κράτη-μέλη που επιθυμούν να επανέλθουν στη ημερινή ώρα μπορούν να το πράξουν αυτό την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Εντάξει. Ε, με βάση την επικουρικότητα τα κράτη-μέλη ε, θα αποφασίσουν μόνα τους αν θέλουν να έχουν ε, μόνιμη θερινή ή χειμερινή ώρα η απόφαση για την στάνταρτ ώρα. Αυτό ήταν πάντα εθνική αρμοδιότητα. Όμως για να υπάρχει συντονισμένη προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να διαβουλευτούν πριν καταλήξουν. Γιατί αν κάθε κράτος τώρα έχει διαφορετική ώρα αυτό δεν είναι καλό. Και εμείς προτείνουμε και ένα νέο σύστημα όπου ένα κράτος μέλος που θέλει να κάνει και άλλες περαιτέρω αλλαγές στη standard ώρα στο μέλλον να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποφασή του τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν προκύψει αλλαγή. Έτσι ώστε και άλλα κρατη κράτη-μέλη και οι ενδιαφερόμενοι να είναι ενημερωμένοι. Και τέλος, όσον αφορά τον, ε, την πρότασή μας, ε, τα κράτη-μέλη είχαν ήδη επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων ε, το φθινόπωρο και το αποτέλεσμα θα αναφέρεται σε μια έκθεση πρόοδου που θα κατατεθεί ε, στις 31 ε, Δεκεμβρίου. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι ε, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα καλό χρονοδιάγραμμα, να υπάρξει συμφωνία στην πρότασή μας έτσι ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι άλλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι να έχουν σαφήνεια, να γνωρίζουν τι θα γίνει. Βεβαίως έχουμε ενημερωθεί για τον προγραμματισμό σας που λέει ότι το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους. Εμείς θα θέλαμε η συμφωνία ή ε, δυνατόν να προκύψει νωρίτερα έτσι ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω στις ερωτήσεις σας και στη συνεργασία μαζί σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά δεν μας είπατε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για αυτή τη στιγμή. Για πείτε μας. Η θέση του Συμβουλίου θα εκφραστεί από το Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου. Δεν εξαρτάται από μένα να εκφράσω εγώ το Συμβούλιο. Si vous avez des informations, vous pouvez nous αν έχετε πάντως πληροφορίες, θα μείνω μεταξύ μας, να το ξέρετε. Il y a personne de la commission qui veut nous donner des infos. Ok, on continue. Madame la rapporteure. Kiria, ici, Kiria. Est-ce que Tack för ordförande och tack för informationen från kommissionen. Karisto, Ίσως να μην ε, κάλυψε όλες τις αμφιβολίες που είχαμε η Κομισιόν. Ίσως να μην ε, Τη δώσαμε αρκετά κίνητρα για να μας δώσει όλες τις απαντήσεις. Εμείς είχαμε ζητήσει πάντως να κάνει μια ανάλυση των ε, συνεπειών αυτής ε, της ε, κατάργησης της αλλαγής της ώρας. Η Κομισιόν τι έκανε στη διάρκεια του καλοκαιριού συνέταξε την πρόταση και μας την υπέβαλε το Σεπτέμβριο και είδαμε πως αυτή η διαδικασία ήταν πολύ γρήγορη και ίσως να μην ε, μπήκε σε, ε, στο απαραίτητο βάθος ή εν πάση περιπτώσει στις λεπτομέρειες που εμείς θα θέλαμε. Ελπίζουμε πως αυτή η πρόταση δεν θα περιπλέξει τα πράγματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εμείς δεν θα το αφήσουμε. Θα συνεχίσουμε να έχουμε υψηλές ε, προδοκίες και φιλοδοξίες και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε ε, πληροφορίες κλειδί, κλειδιά και σαφείς αναλύσεις για την εναλλακτική ε, όσον αφορά την αλλαγή της ώρας. Εύχομαι λοιπόν να μπορέσουμε να μπορέσει μάλλον να υποστηριχτεί αυτή η πρόταση και από πλευρά του Κοινοβουλίου και φυσικά θα πρέπει να δουλέψουμε πιο εντατικά ώστε να ολοκληρωθεί το θέμα πριν το τέλος της θητείας. Ε, τώρα, ποια είναι η ώρα η επίσημη και ποια είναι η ηλιακή ώρα. Αυτό το θέμα απασχολεί πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Ε, κάθε χρόνο έχουμε ε, λαμβάνουμε μάλλον μέτρητα γράμματα από πολίτες που ενδιαφέρονται, μας ζητούν να παρέμβουμε και περιμένουν να υποβάλουμε και προτάσεις δίκες. Εγώ λοιπόν είχα πολλές επαφές με ένα σωρό πολίτες που μου είπαν ότι αισθάνονται άσχημα κάθε φορά που αλλάζει η ώρα. Υπάρχει δηλαδή και θέμα υγείας για πολύ κόσμο. Και αυτό προκύπτει και από την περιγραφή της Κομισιόν που διαπίστωσε την ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Είναι λοιπόν σημαντικό για όλους να υπάρξει ένα εναρμονισμένο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εσωτερική αγορά η οποία εξαρτάται από μία δομή που να είναι προβλέψιμη όσον αφορά τα ωράρια και τις ε, ε, ζώνες ε, αλλαγής της ώρας. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα λειτουργικό, αποτελεσματικό. Με τους σκιώδεις συζητητές έχουμε ήδη οργανωθεί ώστε να προετοιμάσουμε τις επόμενες συνεδριάσεις και να εργαστούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να λάβουν τις ε, πληροφορίες από πλευράς μας. Κανονικά θα έχουμε και μια κατάλληλη μεταβατική περίοδο, αλλά και χρόνο για να προετοιμαστεί το νέο σύστημα. Πρέπει να απλοποιήσουμε τη ζωή των πολιτών λοιπόν και όχι να την περιπλέξουμε ακόμη περισσότερο. Εγώ λοιπόν θα εργαστώ με όσο γίνεται πιο φιλόδοξο τρόπο ώστε να εγκριθεί η έκθεση εντός του τέλους του χρόνου. Θα συνεργαστώ φυσικά με τις επιτροπές που δεσμεύονται για, ε, και εργάζονται για αυτά τα θέματα. Θα συνεργαστώ και με όλους τους κοιόδες με τους οποίους είχα ήδη άτυπες ε, επαφές. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση με τους ε, ε, σκιώδης ώστε να αρχίσουμε τη δουλειά μας και να ολοκληρώσουμε και τη δουλειά μας όσο γίνεται πιο σύντομα μέχρι τα τέλη του έτους. Μέχρι τα τέλη, μάλλον, συγγνώμη, της θητείας. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια. Κύριε Μπόντα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για τα όσα ακούσαμε από την Κομισιόν. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η πολιτική ευελιξία εγώ ηγήθηκα μιας άτυπη ομάδα εργασίας ε, για τέσσερα χρόνια και ασχοληθήκαμε με ένα σωρό τέτοια θέματα. Στι αρχές λάβαμε μια επιστολή ε, από την αρμόδια επίτροπο που έλεγε ότι αυτό το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη τη, αλλά στην έκθεση για την κατάσταση της Ένωσης ακούσαμε από τον κύριο Γιούνκερ πως είναι σημαντικό το θέμα και μάλιστα η Κομισιόν επέβαλε την πρότασή της χωρίς αντίκτυπο, χωρίς μελέτη αντικτύπου. Δεν έκανε δηλαδή αυτό που ζητάει το Κοινοβούλιο και ήμασταν παρόντες σε πολλές συζητήσεις που αφορούσαν τις τη διοργανική συμφωνία όπου αναφέρονται μελέτες αντικτύπου εξάντε και εξπόστ. Βλέπουμε όμως ότι εδώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Καμία απολύτως μελέτη αντικτύπου δεν έχει γίνει. Η δημόσια κρόαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια μελέτη αντικτύπου. Δεν αρκεί. δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο οι εταιρείε μεταφορών θα μπορέσουν να δεχτούν και να ανταποκριθούν σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, γιατί εκείνοι χρειάζεται να προγραμματίσουν εκ των προτέρων. Οι ε, ε, εταιρείε ε, των υπολογιστών θα έχουν δυσκολίες επίσης, γιατί και εκείνοι πρέπει να ε, φτιάξουν προγράμματα υπολογιστών τα οποία θα επηρεάσουν τις αλλαγές αυτές. Κανονικά έχουμε ένα πρόγραμμα διετίας για την εφαρμογή της οδηγίας, ενώ εδώ έχουμε μόνο λίγους μήνες. Ε, πραγματικά δηλαδή θα πρέπει αυτά όλα να εφαρμοστούν σε χρόνο ρεκόρ και δεν έχουμε μελέτη αντικτύπου επί της οποίας να βασίσουμε την εργασία μας. Ένα πράγμα είναι ε, εμφανές, ότι δηλαδή οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θέλουν να ε, καταργηθεί η αλλαγή της ώρας. Τώρα δηλαδή εξαρτάται από εμά να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να το εφαρμόσουμε. Όσο γίνεται πιο γρήγορα, τουλάχιστον αυτό νομίζω μπορούμε να το καταφέρουμε. Ευχαριστώ κύριο Λοτόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, δεν θέλω ε, να πάρω θέση υπέρ ή κατά τη πρόταση. όπου όμως θα πρέπει να θέσω ορισμένα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινώ λοιπόν. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο. Δύο φορέ το χρόνο λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά όλοι στην Ευρώπη έχουμε μέρα και νύχτα περίπου τις ίδιες ώρες. Μετά την αλλαγή μπορεί από τις ε, Βρυξέλλες για να πάει κανείς στο Στρασβούργο να αλλάξει ε, ζώνη, ε, χρονική ζώνη δύο φορές. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Επιπλέον έχουμε προβλέψει ένα χρονοδιάγραμμα που είναι αρκετά στενό. Την επόμενη άνοιξη πολλές επιχειρήσεις μπορεί να μην είναι σε θέση να το πράξουν αυτό ή να πληρώσουν μεγάλο τίμημα για την υλοποίηση μιας ε, τόσο ταχείας διαδικασίας. Έχετε εξετάσει τις συνέπειες ε, αυτής της απόφασης, για παράδειγμα για τις ε, αεροπορικές εταιρείες, γιατί προβλέπει αυτό πολύ μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις χρονικές θηρίδες, τα time slots για τα αεροπορικά ταξίδια. Για παράδειγμα, όταν αλλάζει η ώρα υπάρχει αυξημένος αριθμός ατυχημάτων, ακούω. Υπάρχει, υπάρχουν και άλλα τέτοια επιχειρήματα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτή την απόφαση. Και περιμένω, παρακαλώ, τις απαντήσεις σας. ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το θετικό σε αυτή την πρόταση, ότι δηλαδή χάρη στη συζήτηση στην Κομισιόν και τις προθέσεις της Κομισιόν, μια δημόσια διαβούλευση έχει γίνει, δόθηκαν τα στοιχεία και μαζικά ο κόσμος ε, εκφράστηκε προς μια κατεύθυνση και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας ευχαριστήσει γιατί ήταν το πρώτο βήμα. Δεύτερον, ε, επίση κατέστη σαφέ ότι οι ιστορικοί λόγοι που, στο οποίο οφείλονται αυτές οι αλλαγές της ώρας Η ενεργειακή κρίση δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ισχύει πια, οπότε ε, δεν δικαιολογούνται ίσως αυτές οι αιτήσιες αλλαγές. Και έπειτα υπάρχουν διάφορες μελέτες, ε, αν και δεν είναι και τελείως ε, οριστικά τα πορίσματα, ότι επηρεάζουν τους ανθρώπινους βιορυθμούς και τη φύση αυτές οι αλλαγές της ώρας. Αν και όπως είπα δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς όλα αυτά. Τουλάχιστον λοιπόν πρέπει να το σκεφτούμε. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια απόφαση σε σχέση με το θέμα αυτό. Όμως υπάρχει κάτι που μας ανησυχεί πραγματικά. Αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι άλλο είναι να μην γίνεται αυτή η εποχική αλλαγή δύο φορές το χρόνο, θα πρέπει να αυτό να σταματήσει, αλλά και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποια ε, ε, επίσημη ώρα θα τηρήσουν γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια και ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη ώστε να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις τους διότι προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε εναρμονισμένη ε, εστίαση σε αυτό το θέμα, εσωτερική συνοχή και ανάλογα με το τι κάνουν τα κράτη μπορεί να υπάρξει τεράστια στρέβλωση σε όλους τους τομείς ε, μπορεί να επηρεαστεί λοιπόν η ευημερία των, ανθρώπων. Ε, μην ξεχνάτε την ε, αεροπορία. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με βάρδιες, μέρες, νύχτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε με αυτή την ανησυχία είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε και αν θεωρούμε πως δεν ισχύουν πια ιστορικοί λόγοι στους οποίους οφείλεται η αλλαγή της ώρας, να σταματήσουμε τις δύο ετήσιες αλλαγές. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιλμπάου. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση βεβαίω και μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές. Ε, τότε είχε εισαχθεί αυτή η ρύθμιση με το αιτιολογικό ότι εξοικονομείται ενέργεια. Αλλά όλε οι έρευνε απέδειξαν ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά γι' αυτό είχε εισαχθεί αυτό το μέτρο. Βεβαίω στην Ευρώπη έχουμε ε, διαφορετικά, ε, διαφορετικές ρυθμίσεις για την ώρα το γεγονός ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν διαφορετική ώρα, ξέρετε που οδήγησε στο ότι ο Χίτλερ, ο Φράνκο και ο Μουσολίνη συνεργάστηκαν και ήθελαν να ρυθμίσουν την ίδια ώρα. Όχι, όχι, κάνετε λάθος, λέει ο κύριος Κράμερ. Κάτι ακούγεται εκτός μικροφώνου, εμείς δεν ακούμε. Όχι, ισχύει αυτό που λέω εγώ. Mm εσείς ε, πάντα πετάγεστε, εγώ θα συνεχίσω να μιλάω. Το γεγονός ότι δεν άλλαξε αυτό μετά το πόλεμο δεν το καταλαβαίνω, αλλά τώρα υπάρχει μια κατάσταση όπου έχουμε ζώνες ώρας και ξέρουμε ότι αυτό είναι βλαβερό για την υγεία. Ε, τα ζώα ε, και αυτά έχουν πρόβλημα. Δεν ξυπνάνε με το ξυπνητήρι, αλλά έχουν πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας. Βεβαίως και υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Στο βορρά υπάρχουν άλλα συμφέροντα από ότι στο νότο και ίσως και στη δύση. Αλλά βεβαίως εμείς δεν θέλουμε ένα μπαλωμένο πράγμα. Θέλουμε να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ανεκτό ε, και θέλουμε να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας γιατί σήμερα πλέον δεν φέρνει κανένα προτέρημα, κανένα πλεονέκτημα. Η κυρία Κιόνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. για τη δουλειά που έχει κάνει, για τους Φινλανδούς. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Εδώ και πολύ καιρό μας απασχολεί. Ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο Σβόποντα για την ε, πολύ καλή συνεργασία μέχρι τώρα. αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Οι εμπειρογνώμονες αυτή τη στιγμή ε, εστιάζουν τον προβληματισμό τους στις μεταφορές, ιδίως στις αερομεταφορές. Και ήθελα να επισημάνω ότι όταν εξετάσουμε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Πώς θα γίνει ο επαναπραγματισμός του χρονοδιαγράμματος των ε, αεροπορικών ε, μεταφορών. Αυτό θα πάρει χρόνο και πρέπει να υπάρξει και σημαντική διαβούλευση και διαπραγμάτευση. Γι' αυτό και ελπίζω να υπάρξει πανευρωπαϊκή λύση για να μην έχουμε πολύ διαφορετικές ε, χρονικές ζώνες και λύσεις. Και αυτό να δημιουργήσει από μόνο του πρόβλημα για όλο το σύστημα μεταφορών, ιδίως τις αερομεταφορές αυτό. Ελπίζω λοιπόν να είμαστε σε θέση να αφήσουμε πίσω μας αυτή την ε, αλλαγή ώρας ε, κάθε λίγο και λιγάκι, χωρίς όμως ε, να υπάρξει κατακαιρματισμός των χρονικών ζωνών και έτσι να έχουμε μια χειρότερη κατάσταση από ό,τι έχουμε σήμερα. Να βρούμε λοιπόν μια λύση για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κιλόνεν. Κυρία Αγναουτσού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούγκερ επισήμως ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι δεν ε, θα χαρούν αν εμείς συνεχίσουμε να αλλάζουμε την ώρα κάθε δυο, κάθε εξάμενο μάλλον. Και τώρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν από μόνο τους αν οι πολίτες τους ε, θα ζουν ε, με τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Τέλος παράθεσης. Τώρα, ξαφνικά έχει γίνει κάτι το κατεπήγον το θέμα της ώρας. Δίνει λοιπόν αυτό την εντύπωση και εν ώψη και των ευρωεκλογών ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει τους πολίτες, ότι η Βρυξέλλες δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική μηχανή ε, και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκδηλώσουν τις απόψεις τους μέχρι τον Απρίλιο. Για να αποφύγουμε όμως ε, μια εμβαλωματική προσέγγιση, οι κυβερνήσει θα πρέπει να συμφωνήσουν. Οι νότιοι πληθυσμοί προτιμούν τη θερινή ώρα, οι υπόλοιποι τη χειμερινή. Και τώρα πού να πάμε και στις απόψεις ε, των ε, επιμέρους κλάδων. Ήδη οι αεροπορικές μεταφορές ζητούν τουλάχιστον 18 μήνες χρονικό περιθώριο. Ο καθένα λοιπόν λέει τη δική του γνώμη, ακόμα και στι μεγάλε πολιτικέ ομάδε δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Εγώ τίνω προ τη θερινή ώρα, άλλοι θέλουν την ε, χειμερινή. Και βλέπουμε ότι και στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν έχουμε ανατολή την ίδια στιγμή ανάλογα με την περιοχή που βρισκόμαστε. Επομένω, με αυτό το πρόγραμμα μήπω δημιουργούμε προβλήματα που μέχρι τώρα δεν υπήρχαμε, έτσι αναφέρει ειρωνικά ένας ε, υψηλά ειστάμενο ε, υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει λάβει υπόψη το βασικό πρόβλημα των Ευρωπαίων σήμερα ενώπιση των εκλογών που είναι η ανεργία. Δεν νομίζω τώρα ότι οι φτωχοί και οι άνεργοι θα ευχαριστήσουν τον Γιούνκερ ακόμα και σταματήσει η αλλαγή τη ώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Ντέλε, έχετε το λόγο. Για ένα λεπτό. Ενάμιση λεπτό. Εντάξει, συντομία λοιπόν. Είναι φυσικά ένα μεγάλο δίλημα και ο δημόσιος διάλογος που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ εντυπωσιακό, με συμμετοχή 4,6 εκατομμυρίων πολιτών. Αν δείτε όμως ε, την πρόταση της ε, Κομισιόν, δεν βλέπω κάποιο μέσο επίτευξης ε, του στόχου της ενιαίας λύσης. Γιατί τελικά εδώ πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ δύο βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικουρικότητα, δηλαδή διαλέγουν τα κρατημέλη, και ενιαία αγορά από την άλλη. Εναρμονισμένοι κανόνες. Το πρόβλημα λοιπόν πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από ό,τι φαίνεται εκ πρώτη όψης. Και καταλαβαίνω ότι σιγή του Συμβουλίου. Δεν βλέπω κάποια διέξοδο, κάποιον τρόπο συμφιλίωσης αυτών των αντίθετων ε, αρχών στο ίδιο έγγραφο, στην ίδια οδηγία. Αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση μπορεί να έχουμε ακόμα περισσότερες ε, διχογνωμίες και πραγματικά πρέπει να πω ότι δεν είναι αυτή η σωστή στιγμή για κάτι τέτοιο. Ιστορικά δηλαδή, να, να βρούμε και να ανοίξουμε νέα μέτωπα διχογνωμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Λουκασέντσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εισαγωγή της θερινής ώρας ε, έγινε τον προηγούμενο αιώνα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ε, στο πλαίσιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Μετά είχαμε και την πετρελαϊκή κρίση βέβαια. Σήμερα Έχουμε περισσότερους λόγους για την αλλαγή ώρας, ωστόσο οι Ευρωπαίοι με 5 εκατομμύρια ψήφους έδειξαν ότι επιθυμούν την κατάργηση της αλλαγής της ώρας γιατί δεν συμβάλλει πλέον σε εξοικονόμηση ενέργειας. Και δυστυχώς ε, βλάπτει και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα πρώτα απ' όλα σε ένα τόσο απλό πρόβλημα που είναι η κατάργηση της αλλαγής της ώρας να ακούσουμε τις απόψεις ε, των ψηφοφόρων μας και να ακούσουμε και το βιολογικό μας ρολόι. Να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την πρόταση δεν χρειάζεται να υπάρξουν τόσες αμφιβολίες. Αυτοί που μίλησαν προηγουμένως ε, για τα ωράρια και τις χρονικές θηρίδες των αερομεταφορών. Μπορεί να υπάρχουν τέτοια ζητήματα, αλλά θα λυθούν αρκετά εύκολα, πιστεύω. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένη ότι πρέπει πραγματικά να ακούσουμε τις προθέσεις των πολιτών μας και να ακολουθήσουμε την κοινή λογική για να άρουμε τις ε, επιζήμιες προεκτάσεις της αλλαγής της ώρας. Η κυρία Αγιάλα Σαντέρ. Eh, Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν ε, γιατί για μένα ήταν έκπληξη και μου Ήρθαν κάποια απορίες για το πώς αξιολογείται τη σύγκριση ανάμεσα σε αυτό το είδος τη διαβούλευση και την αντίδραση, την άμεση αντίδραση της Κομισιόν, ενώ όταν πρόκειται για πρωτοβουλίες του πολίτη, απαιτείται να τηρηθούν πολύ περισσότερα κριτήρια για να τα υιοθετήσει ως πρωτοβουλίες η ίδια η Κομισιόν. Σε αυτό το είδος τη διαβούλευση όμως ήταν πολύ πιο άμεση αντίδραση και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη, ώστε στο μέλλον να ζητάμε τέτοιου είδους διαβούλευση αντί για την πρωτοβουλία των πολιτών. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιο αξίζει περισσότερο. Δεύτερο και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Όλξοκ, χρειάζεται εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον πρόκειται για την βελτίωση ε, τον, ε, της κατάστασης τόσο για την, τα ωράρια των, στις μεταφορές όσο και για την ευημερία των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν εναρμόνιση ενώ η επιλογή της ώρας που θα ακολουθηθεί είναι ε, εθνική υπόθεση. Άρα λοιπόν χρησιμεύσε όλο αυτό να βάλουμε ε, ένα θέμα πολύ σημαντικό ε, επιτάπητος, δηλαδή το θέμα της συμφιλίωσης των ωραρίων ε, των οικογενειακών και των εργασιακών. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε και να δούμε πότε θα κλείνουν, πότε θα τελειώνει η εργασία. Θα βοηθήσει λοιπόν αυτό, αυτή η συζήτηση στο να μπορέσουν και οι οικογένειες να συνδυάσουν τα ωράριά σας. Ευχαριστώ κύριο Στεμισμέκερ. Ναι, έχουν ήδη υποθεί πολλά, πολλές παρατηρήσεις έχουν αναφέρει συνάδελφοι και συμφωνώ με την αρχή να φύγουμε από αυτή την ε, αλλαγή κάθε εξάμεινο του χρόνου. 100% υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Όμως, το γεγονός ότι έχουμε προεκλογέ μπροστά μας δεν σημαίνει ότι ξαφνικά πρέπει να βιαστούμε τόσο πολύ και να το σπρώξουμε έτσι στα γρήγορα αυτό το project. Καλή πρόταση, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις ε, δυσμενείς επιπτώσεις για την εσωτερική αγορά που μπορεί να είναι και αρκετά σημαντικές. Γι' αυτό και συμφωνώ με τους αδέλφους που είπαν ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμένη προσέγγιση, οπωσδήποτε γιατί διαφορετικά και για τις μεταφορές, για το εμπόριο, για τον τουρισμό μπορεί να υπάρχουν σημαντικέ προεκτάσεις. Δεν πρέπει να βιαστούμε λοιπόν. Θα ήθελα και ήλπιζα να μας πει κάτι παραπάνω Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Συμβούλιο. Γιατί εγώ από αυτά που ακούω είναι ότι βλέπω ότι δεν προχωρούν οι συζητήσεις εκεί. Υπάρχει ένα κόλλημα. Υπάρχουν πολύ σημαντικέ διαφορές ε, απόψεων και προτιμήσεων μεταξύ Βορρά, Νότου, Δύσης και Ανατολής. Επομένως, η Αυστριακή Προεδρία, να ρωτήσω εγώ, θα αναλάβει βήματα ή το έχει πράξει ήδη εντός του Συμβουλίου και θα προλάβουμε. Merci beaucoup, Monsieur de Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι επιφορτισμένος με το θέμα αυτό από την Επιτροπή Ήτρε ε, και θέλω να σας πω ότι πολλοί συναδελφοί ε, διερωτώνται τι θα κάνουμε αν ε, ορισμένα κράτη-μέλη αποφασίσουν διαφορετικά, κυρίως σε αυτά που είναι γειτονικά κράτη. Αυτό θα είναι τεράστιο πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα της ε, αλλαγής ώρας ε, θα μπορέσουμε να το λύσουμε μόνο αν υπάρχει μηχανισμός ε, συντόνισης ανάμεσα στα κράτη-μέλη που να ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Επ' αυτού θα ήθελα παρακαλώ να έχω μία απάντηση από την Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε ε, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ, κύριε Σινγκριν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Επιτέλους ε, φτάσαμε στη στιγμή που να, μπορούσαμε να μπορούμε να σταματήσουμε δύο φορές το χρόνο να αλλάζουμε την ώρα. Είναι πρόβλημα όχι μόνο για τους κτηνοτρόφους που αρμέγουν τις αγελάδες και είναι σημαντικό αυτό για τις αγελάδες και οι γεωργοί είναι αναγκασμένοι να το μοιράζουν πολλές φορές σε πολλές εβδομάδες αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα και για τα αυτιστικά παιδιά και επίσης και για τους ανθρώπους ε, που έχουν ε, που ε, είναι σε θεραπεία, παίρνουν φάρμακα. Είναι πρόβλημα και για ανθρώπους που διαταράσσεται ο ύπνος τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρείται αυτή η αλλαγή της ώρας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχής με όλο αυτό και θα υπερψηφίσω και ε, για τους ε, καθαρά ε, προσωπικούς λόγους θα πω «Δόξα το Θεό» με το να πρέπει να αλλάξει το ρολόι σε διάφορες συσκευές. Ε, εγώ χρειαζόμουν 9 ώρες για να αλλάξω την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Merci beaucoup, Monsieur Lundgren. Madame Clune, la parole est à vous. Thank you. Σας... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατανοώ τον προβληματισμό, τα ερωτηματικά, λέτε ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμό, να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ε, ζωνών. Το πιο σημαντικό όμω είναι αυτό που ανέφερε ο προηγούμενο ομιλητή. Αν θέλουμε να αλλάζει η ε, ώρα κάθε έξι μήνες ή όχι. Και εδώ υπάρχει συμφωνία. Ότι είναι πρόβλημα να αλλάζουμε κάθε έξι μήνε. Και για τα ζώα, και για τα παιδιά, για όσους έχουν μικρά παιδιά και για τους υπολείπους δηλαδή είναι πρόβλημα. Εάν ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό και συμφωνήσουμε από αυτού, τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Σίγουρα θα καταβάλει τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να υπάρξει συντονισμό κτλ. Ελπίζω να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει ευρύτατη στήριξη για αυτή την πρόταση. Και είναι και φρέσκο γιατί ξαναλάξαμε την ώρα πριν από δυο-τρει εβδομάδες και είδαμε ότι αυτό μας ταράζει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το σκεφτούμε από κοινού και μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και η τεχνολογία σίγουρα θα μας βοηθήσει. Στη χώρα μου υπάρχει μια διαβούλευση αυτή τη στιγμή που λύγει στα τέλη του μήνα και από ό,τι ακούω υπάρχει μια θετική στάση απέναντι στο να σταματήσουμε την αλλαγή της ώρας. Είτε διαλέξουμε τη θετική, θερινή είτε τη χειμερινή ώρα. Κυρία Βερουκίνα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται, συμφωνούμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Σχεδόν όλοι επιδοκιμάζουν την πρόταση, την περιμένουμε από καιρό και βλέπουμε ότι υπάρχει και ευρία στήριξη από τους πολίτες έχουν κουραστεί με την αλλαγή κάθε εξάμεινο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα τώρα να σταματήσουμε αυτό και μάλιστα σύντομα. Από την άλλη υπάρχει και το πρόβλημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να δώσει όλη αυτή την ευελιξία στα κράτη-μέλη. Βέβαια, εννοείται ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δική τους ε, χρονική ζώνη, αλλά δημιουργείται μια σύγχυση σε πολλά κράτη-μέλη στη συζήτηση αν πρέπει να ακολουθήσουν τη χειμερινή ή θερινή ώρα. Και η Επιτροπή λέει ότι απλώς κάποιοι ή μάλλον όλοι πρέπει να μα ενημερώσουν τον Απρίλιο για το τι θα κάνουν. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό. Έχουμε τρει χρονικέ ζώνε στην Ευρώπη και πρέπει να υπάρχει συνοχή και στο μέλλον. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε λοιπόν αυτό έτσι και να έχουμε πολύ διαφορετικές χρονικές ζώνες στα κράτη-μέλη. Απαιτείται λοιπόν συντονισμός. Και η και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει πιο ηγετικό ρόλο. Γιατί ήδη συνεχίζονται δημόσιες διαβουλεύσεις σε διάφορα κράτη-μέλη. Και θα υπάρξει τεράστια σύγχυση αν κάποιος δεν συντονίσει αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε. Μπήκα και εγώ στο κατάλογο μελητών. Να πω και εγώ λοιπόν. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι την πρωτοβουλία, ποιοι την ανέλαβαν, την ανέλαβε η Επιτροπή των Μεταφορών. Αυτή η πρώτη ανέλαβε την πρωτοβουλία ε, για να τεθεί τέλο στην αλλαγή τη ώρα. Δεν είναι λοιπόν πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τη Επιτροπή Μεταφορών. Εδώ και πολλά χρόνια οι Ευρωπαίοι πολίτε μέσω αιτήσεων, μέσω επιστολών έλεγαν ακούστε μας, έχουμε βαρεθεί να αλλάζουμε δύο φορές το χρόνο την ώρα. Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη, ούτε τα κρατη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Μεταφορών έδειξε το θάρρος και είπε ναι λοιπόν θα το θέσουμε σε ψηφοφορία. Αυτό κάναμε τον κύριο Σβόμποντα ε, και είχαμε αυτό το ψήφισμα στην Επιτροπή. Το πρώτο πρέπει να πούμε λοιπόν είναι ότι εδώ και χρόνια δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως είπατε και για την εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Για όσους λένε ότι εντάξει αυτό δεν είναι θέμα προτεραιότητας, προσοχή. Όλες οι μελέτες δείχνουν κάτι που είναι σημαντικό, ότι αυτό θίγει το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Δεν θα κάνω διακρίσεις τώρα ε, για όσου υποφέρουν από αϊπνία και άλλα προβλήματα. Είναι όμως σημαντικά θέματα. 30% του πληθυσμού είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά, εγώ το βλέπω και στη Γαλλία, το θέμα της οδικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της ε, αλλαγής της ώρας, το εξέτασα, γιατί δεν το είχα προσέξει ποτέ. Είδα λοιπόν ότι υπάρχει αύξηση 40% στα ατυχήματα με πεζούς και με ποδηλάτες γιατί δεν υπάρχει φωτισμός και ούτε και η απαραίτητη αντίδραση ενδεχομένως. Λοιπόν, παίρνουμε το θάρρος, το ψηφίζουμε αύριο και ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το περάσει. Υπάρχει όμως ουσιαστικό πρόβλημα. Γιατί κάνετε τη διαβούλευση, όλοι οι πολίτες λένε ναι συμφωνούμε, αλλά δεν εξηγήσατε τη μέθοδο. Κάποια στιγμή είπατε να, θα τα βρουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Μα όχι. Γιατί να δώσετε αυτή την εξουσία στα κράτη-μέλη και να υπάρχει αυτό το θεμελιώδες ερώτημα και πρόβλημα. Είναι ζήτημα ευρωπαϊκής εναρμόνισης η αλλαγή της ώρας. Και τώρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί, πρώτον, με ποιο κριτήριο θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τα κράτη-μέλη αν θέλουν τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Κάθε κράτος μέλος θα κάνει μια δημόσια διαβούλευση. Κυρία Κλούν, εσείς είπατε ότι είχατε δημόσια διαβούλευση στη χώρα σας, έτσι δεν είναι. Ναι, αυτή τη στιγμή γίνεται, μέχρι τα τέλη του μήνα. Και εσείς είπατε. Ναι, αλλά δεν υποχρεωμένα όλα τα κρατη να κάνουν δημόσια διαβούλευση. Υπάρχει λοιπόν έλλειμμα δημοκρατίας από αυτή την άποψη. Εάν σε κάποιες χώρες οι πολίτες μπορούν να εκφέρουν γνώμη και σε άλλες όχι, τι θα γίνει. Πρέπει να ζητήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη να κάνουν διαβούλευση. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Εφιστάτε την προσοχή σας αυτό. η αλλαγή της ώρας είναι εθνική αρμοδιότητα. Το πρόβλημα που, εγώ, έχω εγώ είναι αν δύο γειτονικέ χώρες δεν επιλέξουν την ίδια ώρα. Εγώ είμαι Γαλλίδα, δουλεύω στην ε, Γερμανία. Η μία χώρα έχει θερινή και η άλλη χειμερινή ώρα. Κάθε πρωί και βράδυ αλλάζω το ρολόι μου. Το ίδιο ισχύει και με το Βέλγιο, με την Ιταλία. Τι συμβουλεύω λοιπόν, να γίνει μια ομαδοποίηση των χωρών που θα επιλέξουν την θερινή ή τη χειμερινή ώρα και έτσι θα έχουμε ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Ε, Donc, vous avez vu toutes les questions sur lesquelles on est. Είδατε λοιπόν όλα τα ζητήματα και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να προσέξετε και το είπε και ο κύριος Μάκερ δεν γίνεται να κάνετε εξαγγελίες και να μην τις στηρίσετε. Θέσατε ένα χρονοδιάγραμμα, είπατε 1η Απριλίου όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, δηλώσουν την απόφασή τους. Αυτό τι είναι, αύριο. Και από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα δεν είναι και προτεραιότητα της Αυστριακής Προεδρίας. Βοηθήστε μας λοιπόν και πείτε μας πώς θα γίνει αυτό από τεχνικής άποψης. Γιατί εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εδώ, πολλή νομοθεσία να περάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ πλούσια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστώ μαζί σας γιατί έτσι ε, φαίνεται ότι η Επιτροπή ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ενθαρρυντικό. Πρώτα απ' όλα, κυρία Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Η έκθεση αυτή δεν έρχεται από το πουθενά. Ε, το θέμα αυτό της θερινής ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει στην αντίληψή μας εδώ και αρκετά χρόνια και θέλω να αναγνωρίσω ότι η Επιτροπή αυτή ήταν εκείνη που άνοιξε το δρόμο. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι σε συνδυασμό με τη δική μας πρόταση θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ετέθησαν πάρα πολλά ερωτήματα και κάπως μπορώ να τα κατηγοριοποιήσω. Πρώτον, όσον αφορά το θέμα σχετικά με μελέτη επιπτώσεων, υπάρχει το πολύ σημαντικό θέμα του συντονισμού, δηλαδή πώς μπορούμε να αποφύγουμε ένα ε, εμβαλωματικό σχέδιο για τις ε, χρονικές ζώνες και ποια είναι η θέση των άμεσα ενδιαφερόμενων. Έτσι, και πολύ σημαντικά θέματα σχετικά με την οδηγία ασφάλεια και αυτά δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε. Όσον αφορά στο θέμα της μελέτης αντικτύπου ε, αναθεωρήσαμε, ε, εξετάσαμε τα στοιχεία που υπάρχουν για την ε, θερινή ώρα και σας είπα ότι όλα αυτά ε, αναφέρονται πάρα πολύ ωραία στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Αυτή τη στιγμή ε, τα στοιχεία κατατείνουν σε ένα συμπέρασμα ότι αν δεν υπάρξει συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αυτό θα είναι ιδιαίτερα ζημιογόνο για την κοινή αγορά. Νομίζω συμφωνούμε όλοι από αυτού. Και αυτό μπορεί να προκύψει είτε με τις ε, τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε ε, και με το να γυρίσουν όλοι στην ίδια ώρα. Η κυρία Κλούνη έχει δίκιο, τελικά περί αυτού πρόκειται, πρόκειται για το κατά πόσον θα σταματήσουμε ε, την αλλαγή της ώρας. Δεν πρόκειται για το ποια χρονική ζώνη θα επιλέξουν τα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα σταματήσουμε να αλλάζουμε την ώρα ή όχι. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ήδη εκφράσει την προτίμησή τους ε, στο να σταματήσουμε να αλλάζουμε την ώρα και γι' αυτό ελήφθη μια πολιτική απόφαση. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Πολιτική λοιπόν απόφαση να προτείνουμε την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της κοινή αγοράς, ενώ η απόφαση για το ποια ώρα θα επιλέξουν τα κράτη-μέλη ε, ανάμεσά τους αυτή την απόφαση να την αφήσουμε στα ίδια τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας τομέας όπου πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο. Είναι η κυρίαρχη απόφαση των κρατών μελών να αποφασίσουν μόνα τους ποια χρονική ζώνη θέλουν να εφαρμόσουν. Ε, και αυτό δεν θα αλλάξει με την πρότασή μας. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο ποιες θα είναι μελλοντικέ επιλογές η πρόταση αυτή ε, έχει ως στόχο να προκαλέσει τη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο και είναι αλήθεια ότι αρκετά κρατημέλη ήδη οργανώνουν τις δικές τους τις ε, δημόσιες διαβουλεύσεις. Εμείς ε, αυτό το κρίνουμε ως μια θετική και απόλυτα απαραίτητη εξέλιξη. Τέλος, και εξίσου σημαντικό, αν υποβάλουμε τώρα πρόταση, αν ε, αντιδράσουμε ταχύτατα, τότε αυτό θα είναι σίγουρα θετικό και με τον τρόπο αυτό ε, θα ληφθεί υπόψη και η άποψη της Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά το συντονισμό, αυτή την κατηγορία ερωτημάτων, ο συντονισμός είναι καθοριστική σημασίας. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε να υπάρχει ένα μοσαϊκό διαφορετικών ορών στο μέλλον. Όπως ήδη είπαν τα κράτη-μέλη, έχουμε τρεις χρονικές ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μελλοντικό σενάριο θα εξαρτηθεί από τις επιλογές των κρατών μελών. Πρέπει όμως να είναι απόλυτα σαφές ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν έχουν σχέση με τη θερινή ώρα, έχουν σχέση με την απόφαση των κρατών μελών. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει συντονισμός και έτσι θα είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της κοινή αγοράς. Άρα είναι απολύτως απαραίτητο τα κράτη-μέλη μεταξύ τους να διαβουλευτούν και να συντονιστούν πριν λάβουν τις ε, τελικές τους αποφάσεις. Και μετά ε, θα προτίσουμε σε μία εξέλιξη στο Συμβούλιο και αυτή είναι η ουσία του θέματος. Η Αυστριακή Προεδρία ενδιαφέρεται πάρα πολύ ε, στο να διασφαλίσει το σωστό συντονισμό και εμείς το υποστηρίζουμε αυτόν επιφύλακτα. Όμως ε, πιστεύουμε επίσης ότι αυτή η απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ε, κρατών μελών και ως εκ τούτου συμβαδίζει με τις ευθύνες των κρατών μελών. Εμείς θεωρούμε ότι ο συντονισμός θα πρέπει να γίνει ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου υπό την αγίδα της Αυστριακής μετά της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ε, το ρόλο του διαμεσαλαβητή και θέλουμε να βοηθήσουμε την οποιαδήποτε Προεδρία να καταλήξει σε μια συντονισμένη προσέγγιση πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση στο Συμβούλιο και θα τα συζητήσουμε αυτά και στις 3 ε, Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της έκθεσης πρόοδου ε, στο Συμβούλιο Μεταφορών. Όσον αφορά τώρα τους άμεσα εμπλεκόμενους, αυτό αναφέρθηκε από πολλά μέλη. Βεβαίως και έχουμε δει τα σχόλια ε, των ε, αεροπορικών εταιριών, τις ανησυχίες τους σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της οδηγίας ε, στον επιμερισμό των σλότ και πολλά σχετικά. Το βασικό μήνυμα που παίρνουμε από τους άμεσα ενδιαφερόμενους είναι ότι επιθυμούν να έχουν ένα εναρμονισμένο καθεστώς όσον αφορά την αλλαγή της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν συνέπεια, προβλεψιμότητα και σαφήνεια. Εμείς έχουμε ε, συνειδητοποιήσει ότι η κατάργηση ε, της ε, ώρας, της αλλαγής της ώρας θα συνεπάγεται και κάποιο κόστος για να αποφύγουμε τις αναταραχές. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο έχει συζητηθεί στα κράτη-μέλη, δηλαδή ποιο είναι το απαραίτητο χρονικό διάστημα, το μεταβατικό, για να μπορούν τα κράτη-μέλη να προβούν στη σωστή μετάβαση στην απρόσκοπτη μετάβαση. μετάβαση. Βεβαίως, ε, ε, οι πολίτες ε, δεν αποφελούνται πλέον από το να αλλάζουν την ώρα δύο φορές το χρόνο. Και χαίρομαι που άκουσα τέτοια αμέριστη υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά το θέμα της οδικής ασφάλειας, Βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι. Αυτά που είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις είναι ότι τα στοιχεία για αυτό το συγκεκριμένο θέμα παραμένουν αμφίσιμα όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στη θερινή ώρα και την ε, οδική ασφάλεια. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πότε σκοτεινιάζει και αυτό ε, η οδική ασφάλεια έχει άμεση σχέση με, το, με τη σκοτεινιά. Γιατί όταν σκοτεινιάζει εκεί αυξάνονται οι κίνδυνοι για τροχαία ατυχήματα. Ε, όσον αφορά λοιπόν εμάς, εμείς ε, βασιζόμαστε και σε στοιχεία που υπάρχουν από την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου από το 68 μέχρι το 71. Θεωρούμε ότι τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση ανάμεσα στις θερνές ρυθμίσεις και τα τροχαία ατυχήματα ε, δεν είναι απόλυτα πιστικά, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε με ευαισθησία. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου ε, και προσβλέπω ε, σε μια μελλοντική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για τον ενδιαφέρον σας. Merci beaucoup. La Commission... Και εγώ σα ευχαριστώ, αλλά δεν μα είπατε πώ θα κάνατε για να συντονίσετε το σύνολο των κρατών μελών. Θα σα βοηθήσουμε εμεί. Γι' αυτό φτιάχνουμε αυτή την έκθεση, γι' αυτό είμαστε εδώ και εμεί για να κάνουμε προτάσει και να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα όσα είπε μπροστά στου πολίτε η Κομισιόν αυτή η πρόταση να υιοθετηθεί πριν το τέλο της θητείας. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε με τα μέτρα εξορθολογισμού ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Ο κύριος και δεν ήταν εδώ, δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ, αλλά αντικαθίσταται από τον αγαπητό και μοναδικό Παβέλ Τελίσκα. Ο κύριος Φαντρικά φεύγει μόλις τα από τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε, όπως και ο Ντομινίκ, που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, αλλά βεβαίως μου έδωσε το σημείωμά του. Θα ήθελε λοιπόν να υπογραμμίσει ότι καλωσορίζει την πρόταση της Κομισιόν δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό κανονισμό που θα έχει στόχο να μειώσει το διοικητικό, τους διοικητικούς φραγμούς για τις επενδύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή για την ολοκλήρωση της, των εργασιών στα TNT μέχρι το 2020. Ο εισηγητής θέλει να ευχαριστήσει τους σκιώδες για τις συμβολές τους που σύμφωνα με τον εισηγητή ε, βελτίωσαν ακόμη περισσότερο την έκθεση. Είναι ικανοποιημένο λοιπόν με τη συμβολή των υπολείπων. 180 τροπολογίες. Η πρώτη συνάντηση των σκιωδών ήταν την περασμένη εβδομάδα και εκεί η ε, συνεργασία ήταν θετική κατά τον Ντομινίκρη και οι περισσότεροι σκιώδεις συμφώνησαν για τις κύριες επιτυχίες του κανονισμού να παραθέσω δηλαδή ότι συμφωνούμε για το πεδίο εφαρμογής που θα πρέπει να αφορά τα 10 δίκτυα στον πυρήνα του δικτύου. Επίσης συμφωνήσαμε για μον... Ε, ενιαίες θηρίδες, one-stop shop για κάθε ένα από τα project. Είναι πολύ θετικό ε, που αυτό το ε, την χάνει πολιτικής υποστήριξης. Επίση συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει ένα κράτο μάλλον υπεύθυνο που θα λαμβάνει τελική απόφαση στο τέλος για την ολοκλήρωση του έργου και συμφωνούμε για μια αντιπροσωπεία σε ένα σωστό στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο ανάλογα με το νομικό πλαίσιο του κάθε κράτους από τη στιγμή που τηρείται η αρχή του One Stop Shop και πάλι δηλαδή τονίζουμε αυτό το σημείο να έχουμε τη δυνατότητα ώστε οι αρχές να μπορούν να συντονίζουν τις δράσεις τους, ώστε φτιάχνοντας μια κοινή αρμόδια αρχή για να έχουν πραγματική ορατότητα και πάλι όμως έναν και μόνο συνομιλητή για την ολοκλήρωση του project. Επόμενη συνεδρίαση των σιωδών είναι προγραμματισμένη για το Δεκέμβριο και θα πρέπει να επιτρέψει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και η ψηφοφορία προβλέπεται στις 10 Ιανουαρίου. Να προσθέσω εγώ για τον εαυτό μου ότι Συμφωνώ με τον Ντομινίκ για ένα καλό συντονισμό για μία μόνη ε, θηρίδα για το κάθε project πάνω σε αυτό δουλεύει και η δική μου ομάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάβελ Τελίτκα. Ο κύριος Βιμ Βαντεκάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Τέλιτσκα που μετέφερε τα όσα ήθελε να πει ο συνάδελφος ε, Ντομινίκ Ρικέ. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα μας παρουσίασε ο κύριος Στέλιτσκα, Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο κάναμε την πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών που ήταν επικοδομητική. Ξεχνάω και τη μητρική μου, τα λέω στα αγγλικά. Πολύ χρήσιμη λοιπόν η συνεδρίαση. Πράγματι δεν ακολουθούμε τους ρυθμούς που πρέπει και έχω τρεις παρατηρήσεις αυτή τη στιγμή. Πρώτον, Εάν ορίσουμε μία αρχή, τότε αυτή θα πρέπει να είναι εθνική αρχή. Δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική οργάνωση, περιφερειακή, τοπική ε, ή σε επίπεδο κρατηδίων. Ή μάλλον νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό, αλλά όχι να λέει το α η μία περιφέρεια και το β η άλλη περιφέρεια και μετά τελικά να μην γίνεται τίποτα. Το δεύτερο, σχόλιο της κυρίας Αγιάλα Σέντερ για τις διασυνοριακές αρχές. Γιατί υπάρχει δυνατότητα, για παράδειγμα, στις ιδρομικές γραμμές μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, να έχουμε μια ή να χρειαζόμαστε μια διασυνοριακή αρχή που θα μπορεί και πάλι να ε, δίνει τέτοιες ε, αρμοδιότητες ή να τις αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως ε, εκ μέρους του ΕΛΚ δεν έχω καταθέσει τροπολογίες γιατί νομίζω ότι πολύ γρήγορα ε, και με μεγάλη σαφήνεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση. Εμείς, όπως είναι φυσικό, συμμετέχουμε επικοδομητικά στις συναντήσεις των σκιωδών του κυρίου Ρικέ. και ο Πάβελ ανέφερε προτάσεις που του έχω μεταφέρει προσωπικά. Μέχρι τον Ιανουάριο σίγουρα θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί είναι μεγάλο το διακύβευμα, ιδίω για τα κάτι μέλη, γιατί ε, αν πρόκειται για ε, ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί και χωρίς ε, τις απαραίτητες άδειες, τότε υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες μας στην Επιτροπή Μεταφορών. Καλώς ήρθατε. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Madame Sender, la parole est à vous. Sí, perdón, porque acabo de... Identifico siempre al señor Rique con, con las old times, sorry. yeah. Bien, en este, eh, perdone, que estaba un poco... C'est la coupe de cheveux, au fait, c'est presque pareil. C'est ça, c'est ça, absolument. T'as raison. Bon, eh, sí, quería simplemente eh, agradecer... Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Ερικέ για την εργασία που έχει κάνει και θα πρέπει να Έχουμε υπόψη μας ότι με τόση δουλειά που έχουμε κάνει με τα τέσσερα πακέτα για το σιδηροπακές μεταφορές, το ΣΕΦ1 και το ΣΕΦ2, ακόμα και έτσι λοιπόν, και παρότι έχουμε συντονιστές τόσο πολύ εμπειρογνώμες όπως ε, είναι οι δικοί μας συντονιστές, τόσο ειδικευμένοι. Τελικά αυτό που λείπει πραγματικά είναι διασυνοριακές μονάδες που να μπορούν μέσα από μια συμφωνία που είναι κάπως η ιδέα που είχαμε ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα επικουρικότητας ότι δηλαδή μετά από τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ των κυβερνήσεων για τους διαδρόμους ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρξουν δύο κρατικές μονάδες που θα έχουν ως στόχο να μπορούν να εφαρμόσουν κανονισμούς και νομοθεσίες πέρα από τα ήδη υπάρχοντα. Να μην υπάρχει δηλαδή επικάλυψη κάθε φορά για τις υποχρεώσεις, τις διαβουλεύσεις, τις τεχνικές και τις περιβαλλοντικές μελέτες δηλαδή στο διασυνοριακό τμήμα ε, να μην μπλοκάρονται ε, τα έργα γιατί ακόμα και σήμερα ε, δεν είναι απαραίτητο η εναρμόνιση μεταξύ της διαχείρισης ακόμα και των νομοθεσίας κάθε φορά ανάμεσα στα κράτη όσον αφορά τους διαγωνισμούς, τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, τις μελέτες αντικτύπου, τις μελέτες αντικτύπου στο περιβάλλον. Ελπίζω λοιπόν πως το αύριο θα μπορέσει να ψηφιστεί ήδη για το ΣΕΦ 2021 μέχρι 2027 να μπορέσουμε να εντάξουμε κάπως ένα σπόρο για, αυτές τις, ε, για αυτά τα μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν πάρα πολύ την διασυνοριακή πρόοδο των διαδρόμων. Και επίσης ε, να πούμε και κάτι πέρα των συντονιστών και των συντονιστριών που μέχρι στιγμής έχουν παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, ε, προώθησαν τα projects, ε, έφεραν σε επαφή και σε επικοινωνία, μιλούν με τις ε, κυβερνήσεις, Πιστεύουμε λοιπόν πως ο συντονιστής ή η συντονίστρια σε αυτό χρησιμεύει να διευκολύνει, να βοηθήσει, να ανοίξει διάλογο εκεί όπου υπάρχει ε, πάγωμα ή μπλοκάρισμα. Εγώ έχω παρακολουθήσει συνεδριάσεις αυτών των συντονιστών με το πληθυσμό, ας πούμε, στη Βάλτα Όστα. Υπήρχαν πραγματικά πολύ δύσκολα προβλήματα, αλλά εκεί μπόρεσαν να ε, βοηθήσουν. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιου είδους διακρατικές μονάδες για να διευκολύνουν στις διασυνοριακές υποθέσεις. Ευχαριστώ. Euh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ, όπως σας έχω ήδη διευκρινίσει, η ομάδα μου είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική. Το είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση και αυτός ο σκεπτικισμός αφορά και το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ρίκε, αλλά και τα ίδια τα project. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τεθούν σε εφαρμογή αυτού του είδους τα project σε πολλά κράτη όπου οι αρμοδιότητες των τοπικών αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπλέκονται ή επικαλύπτονται και η δημιουργία συντονιστικών μονάδων θα ήταν χάσιμο χρόνο. Εάν δεν υπάρξει ταυτόχρονα και η κατάργηση των παλαιότερων δομών για κάθε project. Πρέπει να δούμε δηλαδή τι γίνεται με το χώρο, τι γίνεται με το περιβάλλον, τι γίνεται με ε, το περιβάλλον. Οπότε μια μόνη διαδικασία, μια μόνη ομάδα θα μπορούσε να υλοποιήσει όλο αυτό όλες αυτές τις πτυχές και να εξετάσει όλες αυτές τις πτυχές. Άσε δε που ο χρόνος που θα χρειαζόταν για κάτι τέτοιο θα ήταν ε, απροσμέτρητος. Για τα project κλειδιά λοιπόν, για τα θέματα αυτά της, ε, ε, των υποδομών, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι συνεπή με τον κανονισμό. Να αναπροσαρμοστεί αυτή η διαδικασία ώστε να μπορέσει να ε, συμμορφωθεί προς την νομοθεσία που ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη. Η πρότασή μας λοιπόν θα βασιστεί στη λήψη υπόψη αυτών των διαφόρων τροπολογιών που προτείνουμε στην τελική εκδοχή, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε την υποστήριξή μας όπως έχουν τώρα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, και τον εισηγητή και τη συνεργασία και για τη συνεργασία που μόλις τώρα ξεκίνησε. Νομίζω λοιπόν ότι από τα λάθη μας θα πρέπει να μαθαίνουμε οι διασυνοριακές συνδέσεις Βεβαίω και πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας. Έχουμε την κατάσταση όπου η Ισπανία τότε έφτιαξε έναν αυτοκινητόδρομο στα Πυρηναία τον πήγε μέχρι τα σύνορα και μετά είπαν οι Γάλλοι, όχι, εμεί δεν το συνεχίζουμε. Και ξέρετε τι γίνεται, αυτό ο αυτοκινητόδρομο καταλήγει σε ένα χωριό. Μα αυτό είναι σπατάλι χρημάτων. Ή στη Γερμανία αυτή τη στιγμή συζητάνε τον αυτοκινητόδρομο να ε, τον ε, εξοπλίσουν ε, με ηλεκτρικό ρεύμα αλλά αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με τους σιδηρόδρομους. Όσο και αν είναι ωραίο το ότι υπάρχουν εθνικοί φορείς και εδώ έχουμε εμπειρία. Παραδείγματο χάρη στα γερμανικά-πολωνικά σύνορα. Εκεί υπήρχαν δύο αρχέ που συνεργάζονταν και ήθελαν να κάνουν διασυνορικά προγράμματα. Το πήρε χαμπάρι η πολωνική κυβέρνηση και είπε Μπα, όχι, αυτό είναι δικό μα καθήκον. Αυτό είναι εθνικό θέμα, δεν είναι διασυνοριακό. Το σταμάτησαν λοιπόν αυτό το έργο και δεν συνεχίστηκε γιατί αυτοί δεν έχουν ιδέα. Είναι ώρα λοιπόν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανεί να έχει μία συνταγή. Αν πει κανεί εδώ στο Βέλγιο ότι η Μαντί και η Βαλόνη ε, είναι υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης, θα υπάρξει επανάσταση αν το πει κανεί αυτό. Ε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Βεβαίως και θέλουμε να υπάρχει δίκαιη νομοθεσία. Δεν θέλουμε κυρίως να μειώσουμε τους ε, σιδηρόδρομους. Θέλουμε διαφάνεια που δεν υπάρχει πάντα. Ας πούμε μεταξύ Λιών και του Τωρίνου όλο αυτό το έργο για πόσο καιρό δεν είχαμε ενημερώσει ενημέρωση και μετά θέλουμε να εξασφαλίσουμε και τη συμμετοχή των πολιτών. Μερικές φορές είναι χρονοβόρα η διαδικασία, άλλες ε, πάλι φορές, παραδείγματο χάρη η διαδρομή στην κοιλάδα του Ρήνου κράτησε 20 χρόνια γιατί είχαν πει ότι οι πολίτες δεν έχουν λόγο. Αν τους είχε κανείς συμπεριλάβει από την αρχή δεν θα χρειαζόντουσαν 20 χρόνια. Και βεβαίως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι νόμοι για το περιβάλλον. Παράδειγμα, στην ε, αυτοκινητόδρομο στην Πολωνία έπρεπε να κατασκευαστεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Ευτυχώς δεν κατασκευάστηκε και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όλα αυτά πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κιλόνεν, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Αγαπητέ, τι πρόεδρε, συνάδελφοι. Και για μένα αυτή η πρόταση με αυτό το one-stop shop δεν ε, ήταν πολύ σπουδαία ιδέα. Και το πρόβλημα έχει να κάνει και με το συνταγματικό δίκαιο. Επίσης νομίζω ότι μπορούμε να επιμείνουμε όσον αφορά το ρόλο των κρατών μελών, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα που είναι υπαρκτά. Και ξέρουμε ότι τέτοιου είδους project, τέτοιου μεγέθους, εν γέννη χρειάζονται και ε, τα κτλ. Και αυτά είναι πράγματα που χρειάζεται να αποφασιστούν έγκαιρα και για τη χρήση της γης, ίσως ε, ε, και η χωροταξία είναι αποκλειστική η αρμοδιότητα των Δήμων κανονικά και δεν μπορεί εκεί να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, αυτό που προτείνει η Κομισιόν ε, να εκδίδονται δηλαδή όλες οι άδειες σχετικά με κάθε project από μόνο μία ρυθμιστική αρχή, η ιδέα είναι ε, υπέροχη. Λιγότερη γραφειοκρατία, μόνο μία θηρίδα, ταχύτερη διεκπαιρέωση, όμως είναι μια ριζική αλλαγή όσον αφορά τις αρμοδιότητες των αρχών που εμπλέκονται σε τέτοια project. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι δυνατόν από την άποψη του συντάγματος και επίσης ε, το κάθε κράτος ορίζει την αρμόδια αρχή ανάλογα με την νομοθεσία του πράγμα το οποίο παίρνει χρόνο αν θέλουμε να τα αλλάξουμε. Ο, καθώς και η δεσμευτική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί και θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές άδειες ε, απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί από μία αρχή την οποία ορίζει ο νόμος. Στη συνέχεια αυτό θα πρέπει να επιβληθεί σε εθνικό επίπεδο και ως εκ τούτου προκύπτει ότι έχουμε προβλήματα με το συνταγματικό μας δίκαιο εάν ορίζουμε κάποια διαφορετική αρχή που θα πρέπει να αποφασίσει για το είδος της ε, ζώνης για, κάθε, για, τέτοια project. Σύγκρουση λοιπόν με το Σύνταγμα. Όταν είναι απαραίτητη η εισαγωγή νόμου ε, για το σχεδιασμό, τη χωροταξία που μπορεί να μεταφερθεί από το Δήμο ίσως ε, στο κρατικό επίπεδο. Ίσως ε, να είμαι ήδη πολύ καιρό στην πολιτική. Εγώ πάντως δεν θα βιαζόμουν να προτείνω κάτι τέτοιο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δεν είναι εύκολο. Το είπα στους συναδέλφους και στην ε, συνεδρίασή μας και έδωσα το μήνυμα στον Ρικέ γι' αυτό ότι ευχαρίστω ε, να είχαμε ένα συντονιστικό ρόλο μιας, ε, ενός γραφείου εάν αυτό συμφωνούσε με το Σύνταγμα αλλά αν θέλετε να προχωρήσουμε έτσι, χωρίς να λέμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποιος ρόλος για τους Δήμους και τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές Χωροταξίας και Πολεοδομίας, μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Τώρα όμως δεν λέμε με την πρόταση του ΡΙΚΕ κάτι τέτοιο και αυτό με ανησυχεί. Βεβαίω, αν άλλοι είναι έτοιμοι να καταπατήσουν το συνταγματικό τους δίκαιο, οκ, okay, εγώ τουλάχιστον το δηλώνω και γι' αυτό το λόγο δεν ύψωσα ακόμα την πράσινη σημαία Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με το θέμα αυτό του συνταγματικού δικαίου και ίσως εσείς να μπορέσετε να μας καλύψετε και να καταλάβετε την προβληματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κιλόνεν. Ήμουν στη συνάντηση των σκιωδών όπου εξηγήσατε τους προβληματισμούς σας. Τα γνωρίζουμε λοιπόν. Τώρα, Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Βερζίνη. Παρακαλώ. DG Move. Merci beaucoup, Monsieur le Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τον ε, κύριο Τέλιτσκα που παρουσίασε ε, την πορεία της συζήτησης. Με τα χαρά σημειώνω ότι οι εργασίες στο Κοινοβούλιο ε, προχωρούν αρκετά γρήγορα και επικοδομητικά. Όπως ανέφερε ο κύριος Τέλιτσκα, αρκετά σημεία ήδη ε, αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Ευρωβουλευτών και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Κάτι που αναφέρθηκε και εισαγωγικά από τον εισηγητή είναι ότι αυτή είναι μια σημαντική πρόταση στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου για την κινητικότητα, όμως θα πρέπει να το δούμε και σαν ένα επιπλέον εργαλείο ε, για να υλοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών εν ευθέτω χρόνο και αυτό μαζί και με το MIE2, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή και θα υποβληθεί σε ψηφοφορία αρκετά σύντομα. Σε αυτό το μικρό χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι υπάρχει ευρία στήριξη για την πρόταση. Υπάρχει βέβαια μια σειρά τροπολογιών για την ενίσχυση του ε, κειμένου, για να το βελτιώσει και για να βελτιώσει και το επίπεδο φιλοδοξίας. Με ενδιαφέρουσες προτάσεις ε, για την διασύνδεση της ε, πρόταση αυτή. με άλλα ε, εργαλεία που έχουμε προτείνει. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Έχουν δυνατότητα να δώσουμε, κάνουμε κάποιε διευκρινήσει για μια σειρά πράγματα. Τώρα, πρώτον, το πεδίο εφαρμογή που αναφέρθηκε. Είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα πεδίο εφαρμογή για το κεντρικό ε, δίκτυο TNT, οι διασυνοριακές ε, μεταφορές είναι πολύ σημαντικές και ε, έχουν πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουν, όμως και τα εθνικά τμήματα των διασυνοριακών μεταφορών είναι πολύ σημαντικά πολλές φορές. Γι' αυτό και εμείς ε, θέλουμε να επικεντρωθούμε στο κεντρικό δίκτυο. Άλλο σημείο που συζητείτε είναι αυτό της ενιαίας αρμόδιας αρχής. να έχουμε δηλαδή έναν πιλότο στη διαδικασία διοδότησης των έργων. Κατά τη γνώμη μας αυτό το μέτρο θα διευκολύνει την υλοποίηση των έργων. Χρειάζεται όμως καλύτερη, καλύτερο συντονισμός και συγχρονισμός ε, της διαδικασίας. Η πρόταση της Κομισιόν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και έτσι θα πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα ανάθεσης ε, της αρμοδιότητας αυτής από την αρμόδια αρχή σε ένα τοπικό υπερφερειακό επίπεδο, αν αυτό αντιστοιχεί και στον ε, χαρακτήρα του έργου. Για να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και συμβατότητα με το εθνικό σύστημα. Τέλος, μία πρόταση που έκαναν πολλά μέλη να προβλέψουμε δομέ στην περίπτωση διαδότησης διασυνοριακών ε, έργων. μα φαίνεται ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Ιδίω τα έργα που είναι δύσκολα, πρέπει να έχουμε κατά νου τη διάκριση μεταξύ του ίδιου του παρόχου ή αναδόχου του έργου, μπορεί να υπάρχει μια επιχείρηση ή κάποια κοινή αρχή, και ε, αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής. Τέλος, για το επίπεδο φιλοδοξίας. Και χρονοδιάγραμμα της πρότασης κανονισμού της Κομισιόν. Υπάρχει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας Θεωρούμε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση και συνάδει πλήρω με το κοινοτικό ενωσιακό δίκαιο και στον τομέα του περιβάλλοντο. Είναι σύντομο το χρονοδιάγραμμα, το κατανοούμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Μπορεί να αποτελέσει δηλαδή πρόκληση η τήρηση του χρονοδιαγράμματος σε συγκεκριμένα σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βερτζίνη. Ο Πάβελ Τελίτσκα για δευτερολογήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα μεταφέρω στον Ντομινίκ Ρικέ το μήνυμα ε, ότι υπάρχει ιδιαίτερα ευρεία στήριξη από τους χεώδεις. Κατανοώ ότι υπάρχουν ορισμένα λίγο πιο δύσκολα ζητήματα. Πρώτον, για την ενιαία αρμόδια αρχή Φυσικά και δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του Ντομινίκ Ρικέ. Όμως, εγώ το βλέπω σαν μια διαδικασία. Αν δείτε τι θα ψηφίσουμε αύριο, Μπορεί να μην έχουμε όλα όσα έχουμε εδώ σε αυτό το φάκελο, αλλά η ίδια η ενιαία αρμόδια αρχή θα έχει την πρόθεση να υλοποιήσει τον ε, συντονισμό. Πρέπει να το προσπαθήσουμε. γιατί εν μέρη καθυστερούμε και δεν αποδίδουμε ε, πραγματικά, γιατί λείπει αυτός ο συντονισμός. Το γεγονός λοιπόν ότι ο εισηγητής ε, θέλει να κάνει αυτή την προσπάθεια με τη στήριξη των σχεδών είναι θετικό. Εντάξει, υπάρχουν και νομικά ζητήματα, Πρέπει να δούμε πώς αυτό θα αντανακλάται στις συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ εν ολίγης μπορώ να φανταστώ ένα τέτοιο σενάριο, αλλά θα δούμε τι θα πει και ο εισηγητής. Γι' αυτό που είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ. Είναι ένα διαφορετικό ζήτημα υπό την ίδια κατηγορία όμως. αντίστοιχη εμπειρία έχουμε και σε άλλους τομείς με τις κοινοπραξίες, για παράδειγμα. Σχεδιασμός, προβλέψεις, εφαρμογή και λειτουργία τους. Και μάλιστα αυτό προέρχεται από τα βορειοανατολικά και από την Πολωνία. Για το θέμα των συντονιστών που ανέφερε η Νές, τολμώ να πω από προσωπική πείρα ότι με τον αριθμό των έργων ο αριθμός των έργων θα ήταν πολύ χαμηλότερος αν δεν είχαμε την συμβολή των συντονιστών. Τέλο πάντων θα μεταφέρω τα όσα είπατε. Στον Ντομινίκ Ρικέ και ευχαριστώ τους Κιώδη. Merci Ευχαριστούμε κύριε Τελίτσικα. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία για αυτή την έκθεση θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου. Συνεχίζουμε. Έκθεση για τροποποίηση της οδηγίας 2008-96 σχέση με τις οδικές υποδομές. Κυρία το έχετε το λόγο. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα του χρονισμού, θέλω να σας πω ότι εδώ και αρκετό καιρό δουλεύουμε για αυτό το θέμα, γιατί προσπαθούμε να σεβαστούμε αυτό που ήταν η ολοκλήρωση και η εφαρμογή του προγράμματος έτσι ώστε να μπορούμε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή στις 3 ε, Δεκεμβρίου. Έγινε η μετάφραση των τροπολογιών πριν από λίγο καιρό και ελπίζω τελικά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να μπορέσουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. και βασίζομαι στην κατανόηση των σχεδόν εισηγητών και των πολιτικών του σωμάτων. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να αναζητήσουμε συμβασμού για να κρατήσουμε και να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά την πρόταση λοιπόν, ε, την αρχική πρόταση, τη γνωρίζετε, είναι μια πρόταση που ε, αφορά κατ' ουσίαν ε, την επεξεργασία της πρότασης της Επιτροπής αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας κατόπιν ε, για να υπάρχει βελτίωση της οδικής ασφάλειας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα επιφανειακά στοιχεία αλλά η πρόταση προτείνει και να ελέγχεται αυτή η ίδια υποδομή. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει προστασία των ευάλωτων ε, κατηγοριών και πέρα από αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προσφέρουμε υποστήριξη στην ε, τεχνολογική πρόοδο, στην ψηφιοποίηση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, γιατί οι ε, δρόμοι που έχουμε κατά νου είναι δρόμοι που αφορούν καθαρά το μέλλον. Όσον αφορά τώρα στις νέες τροπολογίες, τις οποίες έχω καταθέσει, Πρώτα απ' όλα προσπάθησα σε ένα και μόνο άρθρο να συμπεριλάβω τα στοιχεία που αφορούν στον έλεγχο της σταθερότητας της υποδομής και μέσα από τη χρήση των αισθητήρων ε, και τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι μια σημαντική τεχνολογική πρόοδος που κατά την άποψή μου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχω εντάξει στις τροπολογίες είναι η πρόταση να αναλάβουν ευθύνε οι αρχέ, οι οποίε είναι αρμόδιες για την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια. Ε, είτε για την υπάρχουσα υποδομή, είτε για τους νέους δρόμους, είτε και πρόκειται για ξεχωριστά κομμάτια ή άλλα που έχουν συμπεριληφθεί σε νέες υποδομές. Οι ε, συνάδελφοι θα παρουσιάσουν τις ε, τροπολογίες τους και στο τέλος, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε την συνολική επανεξέταση του θέματος. Έχετε λοιπόν το λόγο, αν θέλετε, ο κύριος Δεκάν. Πρόεδρε, και πάλι έχω την μεγάλη τιμή να αντικαθιστώ την κυρία Κλάουδια Σμίτ. Και για να είμαι ειλικρινής, είχα λίγο κουραστεί να μεταφράζω τα κείμενά της από τα αγγλικά στα ολλανδικά, οπότε τώρα θα σας τα πω απλώς ε, στα αγγλικά. Αγαπητοί, κυρία εισηγήτρια, εγώ η κυρία Σμίτ Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε. Τι έγινε, γιατί χασκογελάτε. Serious. Όχι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα σας, παρακαλώ. Λοιπόν, ότι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε ε, για να μειώσουμε το θανάτους στους δρόμους μας. Η οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί κατά πολύ τις περασμένες δεκαετίες και χάρη στις δράσεις της Ένωσης. Ανάμεσα στο 2001 και το 2002 το, ο αριθμός των θανάτων έπεσε στο, κατά 42% και ανάμεσα στο 2010 και το 2016 μειώθηκε και πάλι στο, κατά 90%. Ωστόσο 25.600 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους στους, ανθρώπ, στους ευρωπαϊκούς δρόμους το 2016 παρά τη μείωση και έπειτα μιλάμε για την ευθύνη. Ο κοινό αυτό στόχος δεν σημαίνει απαραίτητο πως η Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό ε, την υπόθεση. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν λάθη και είναι κοινή ευθύνη όλων των φορέων και σε όλα τα επίπεδα να εξασφαλίσουν ότι τα τροχαία ατυχήματα δεν θα οδηγούν, δεν θα ε, καταλήγουν σε ε, θανατηφόρες, ε, θανατηφόρα τραύματα. Γι' αυτό όσο καλά και αν διατυπώσουν οι υπάλληλοι των Βρυξελών το σύστημα του δικτύου, κάποιοι θα εξακολουθήσουν να μεθούν, κάποιοι θα εξακολουθήσουν να κουράζονται ή να κοιτάνε το τηλέφωνό τους ενώ οδηγούν. Οπότε το δίκτυο δεν είναι αυτό το οποίο διατυπώνει τους κανόνες, δεν αρκεί μάλλον να διατυπώνει τους κανόνες, πρέπει και οι πολίτες να τους στηρούν. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Είναι αλήθεια ότι μόνο το 8% των θανατηφόρων τροχαίων γίνονται μέσα στο δίκτυο ε, των πόλεων, γιατί βέβαια στους ε, αυτοκινητοδρόμους δεν υπάρχουν πεζοί, φανάρια κτλ. Πάντοτε οι αυτοκινητόδρομοι θα είναι πιο ασφαλείς από όλου του δρόμου. Εάν θέλουμε να μειώσουμε λοιπόν τα θανατηφόρα τυχαία, θα πρέπει να θαρρύνουμε περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί του αυτοκινητοδρόμου παρά να χρησιμοποιούν το δεύτερο ρεύον δίκτυο. Υπό αυτό το φως η επόμενη ε, η ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα για την Ευρωβινιέτ θα είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια στους δρόμους επίσης. Τελευταία παράγραφος αφορά τη νέα τεχνολογία. Είμαι κατά της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής οδηγίας εν γέννη, αλλά στο ΕΛΚ είμαστε υπέρ της συνεργασίας και της εναρμόνισης των σημάτων και σηματοδοτήσεων των δρόμων, ώστε να επιταχύνουμε την ε, χρήση αυτόνομων ή αυτόματων οχημάτων και φορτηγών. Όσο πιο γρήγορα χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα 3SIN στους δρόμους, τόσο λιγότερα θύματα θα έχουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να συμβάλλουμε στο να δημιουργήσουμε ε, τις κατάλληλες προδιαγραφές. Όμως μόνο ένα αυτόνομο αυτοκίνητο θα λειτουργήσει ασφαλώς, μόνο εφόσον υπάρχει ομοιόμορφη Υπάρχουν ομοιόμορφα στάνταρ για τα σήματα και λειτουργούν υπό συγκεκριμένε συνθήκε. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία μπορεί άμεσα να επηρεάσουν ε, τα σήματα Οπότε ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των αυτόνομων ε, οχημάτων δεν μπορεί να μεταφερθεί στους διαχειριστές των δρόμων. Θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες ε, σύμφωνα με αυτά τα επιχειρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κάμπ και η κυρία Γκράσα Βάντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ε, θέμα, πολύ σημαντικός ο κανονισμός. Θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Βαντεκάμπ. Ελπίζω αυτό που μας διαβάσατε μόλις να μην είναι η γνώμη του ΕΛΚ γιατί υπάρχουν αδυναμίες, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε οι υποδομές να γίνουν όσο γίνεται πιο καλές και ασφαλείς. Δεν μπορούμε απλά να πούμε ότι πάντα οι οδηγοί θα κοιτάζουν το κινητό τους. Μόλις 4% του δικτύου TNT είναι αυτό. Αν δείτε το πρωτογενές οδικό δίκτυο, το 39% των θανατηφόρων ε, ατυχημάτων γίνεται σε αυτούς τους δρόμους. Αν μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση εκεί, εντάξει, αλλά πρέπει να επεκτείνουμε και την προσπάθειά μας και στους υπόλοιπους για να μειώσουμε τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων. Μετά, για τα τούνελ και τις γέφυρες. πρέπει και αυτά να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση οδικής ασφάλειας. Ε, συμβαίνουν πολλά ατυχήματα σε σύραγγες και γέφυρες. Θα πρέπει μετά να συμπεριλάβουμε και τις ε, εξόδου, γιατί και εκεί γίνονται πολλά ατυχήματα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει διακομματική συνένεση ως προς την προστασία των ποδηλατών, ε, των πεζών και των μοτοσυκλετιστών. Πρέπει να υπάρξουν και άλλα μέτρα στην επεξεργασία, παραδείγματο χάρη ε, τα, οι ελάχιστε προδιαγραφές για την οδική σήμανση, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, να υπάρχουν εκθέσεις ελέγχου και να υπάρχει και καλύτερη εκπαίδευση για τους επιθεωρητές. Καλύτερη ενημέρωση και για όσους ε, χρησιμοποιούν και υπάρχουν στις οδικές μεταφορές. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι αυτή η έννοια του self-explaining και self-enforcing rules, αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει σε αυτόν τον τομέα να συμπεριλάβει κατευθυντήριες γραμμές γιατί οι καλύτεροι δρόμοι μπορούν να περιορίσουν τους ε, κινδύνους. Και εξάλλου ε, όλα αυτά ε, μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να εγκρίνουμε καλά και σημαντικά μέτρα. Έχουμε τώρα την, για την Τετάρτη μία συνεδρίαση των σκιωδών και η συγγήτρια είπε ότι είναι ιδιαίτερα ανοιχτή όσον αφορά τις προτάσεις μας. Νομίζω γι' αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ε, δεν πρέπει να βιαστούμε γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε και να δείξουμε κατανόηση για το ότι ενδεχομένως η ψηφορία να πρέπει να αναβληθεί και να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Νομίζω ότι αυτό το οφείλουμε ε, σε όσους ε, πλήττονται και τους αφορά η οδική ασφάλεια. Να κάνουμε πιο γρήγορα, αυτό δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Ο κύριος Ντεμεσ Μέικερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για όλη την ενέργεια και τον ενθουσιασμό της για να ολοκληρωθεί η εν εγκαίρως. Φυσικά και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση από κοινού. Ευχαριστώ και τους αδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Η οδική ασφάλεια με ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους χρήστε του δικού δικτύου, φυσικά και είναι ύψιστη προτεραιότητα και για μα. να επισημάνω τέσσερα σημεία. Πρώτον, Συμφωνώ με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, ούτως ώστε στο μέλλον να αξιολογούνται και να ελέγχονται και οι αυτοκινητόδρομοι. Μετά, είναι σωστή πρόταση να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί για όλο το τμήμα του οδικού δικτύου που χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν θέλουμε δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά χρήματα για να δημιουργηθούν μη ασφαλείς υποδομές. Μετά, σηματοδότηση, πινακίδες, ε, πολύ σημαντικό και ε, κέριο τμήμα του οδικού δικτύου. Ε, ιδίω τώρα που τα οχήματα γίνονται πιο αυτόνομα. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να, θέσει ελάχιστα, να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα σηματοδότησης. Και τέλος, θα ήθελα να προτείνουν στην Επιτροπή μία κοινή μεθοδολογία για τις εθνικές εκθέσεις. Και έτσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιήσουν ε, πιο εύκολα αυτές τις εκθέσεις. Επομένω, περιμένω με ανυπομονησία την επόμενη συνάντηση σκιωδών και προσβλέπω σε συνέχιση της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέλιτσκα και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω και εκπροσωπώ πολλούς συναδέλφους σήμερα. Αυτή τη, στιγμή, αυτή τη φορά εκπροσωπώ τον κύριο Βαν Μίλτεμπιουρ που δεν μπορεί να είναι εδώ λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Ευχαριστεί λοιπόν ε, την εισηγήτρια και τους λοιπούς σκιώδεις για τις τροπολογίες τους. Όμως ε, θα ήθελε να τονίσει ο συνάδελφος ότι εξακολουθεί να στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να επισημάνουν ορισμένες επιφυλάξεις. Με κύρια αυτή που συνδέεται με την πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία πέραν του πεδίου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το σημείο για να μην επιβαρύνουμε τα κράτη-μέλη με επιπλέον διοικητικό άχθος θεωρεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη και τεκμηριωμένη. Βασίζεται ε, σε μεγάλης κλίμακα έρευνα και στοιχεία. Γι' αυτό και θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε φυλακτικοί ως προς την προσθήκη στοιχείων που δεν έχουν ε, διερευνηθεί. Να βασιζόμαστε λοιπόν σε μελέτη τυπού πριν ε, προσθέσουμε κάτι στην έκθεση. Μετά. Τίθεται και θέμα αρχής της επικουρικότητας ε, και αναλογικότητας. Γι' αυτό και πάλι τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το πεδίο εφαρμογή που προτείνει η Κομισιόν. Οι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί είχαν ως στόχο ε, τον περιορισμό του γραφειοκρατικού άχθου για τα κράτη-μέλη και την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Ε, σε ορισμένε περιπτώσει είναι πολύ μεγάλε οι ε, απαιτήσει από τα κράτη-μέλη και υπάρχουν και αλληλεπικαλύψει με διαδικασίε που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι τα κράτη-μέλη θα, θα να εφαρμόσουν την οδηγία, γι' αυτό και θα πρέπει αυτό να είναι εφικτό. Παρόλε αυτέ οι φυλάξει, ε, προσβλέπει σε επικοινωνικέ συνεδριάσει των συντονιστών, συγγνώμη, των σκιωδών ε, και σε ένα θετικό αποτέλεσμα τελικά. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Et je me retourne tout de suite vers la Commission européenne. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στρέφαμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, συγγνώμη. Εδώ ε, είμαι, εκπροσωπώ διάφορους συναδέλφους, αλλά όχι και τον κύριο Κράμερ. Αυτό είναι too much. Υπερβολικό. Όχι, από τον κύριο, τον κύριο Κράμερ δεν τον εκπροσωπώ. Συγγνώμη κύριε Κράμερ, δεν σας είδα. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Προφανώς και υπάρχει διαφορά μεταξύ μας και παρότι γνωριζόμαστε και πολύ καλά εδώ και 15 περίπου χρόνια. Ε, καταρχάς, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αγιούτο, ε, την εισηγήτρια για την πολύ καλή πρότασή της. Ε, το εμείς θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρχουν ε, δυστυχήματα, τροχαία ατυχήματα και επειδή ήταν πολύ καλή η προεργασία, οι προσθήκες που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ λίγες. Ε, δηλαδή θέλουμε εμείς ε, να συμπεριληφθούν περισσότερο στο κείμενο ε, και οι ποδηλάτες που είναι θύματα το 10% των ατυχημάτων είναι με πεζούς και το 40% ε, των ατυχημάτων με ποδηλάτες είναι εκτός των πόλεων. Άρα αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Το είπες και εσύ αυτό. Και βεβαίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση, εκεί δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτό είναι τρελό, γιατί εμείς θέλουμε να στηρίξουμε αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ε, θα επιτευχθεί, αλλά μόνο με προϋποθέσεις. Κατά τα άλλα, επιθυμούμε να υπάρχει καλή συνεργασία και των ε, υπηρεσιών ε, παροχής βοήθειας των ασθενοφόρων γιατί ε, αν είναι κάποια περίπτωση στα σύνορα, θα φύγει το ένα στον φόρο από τη μία χώρα, το άλλο από την άλλη. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Κατ' ουσίαν χρειαζόμαστε συντονισμό στα σύνορα. Αυτό ισχύει για τις σύραγγες, αλλά ισχύει και για τις γέφυρες. Και νομίζω αυτό το παράδειγμα αναφέρθηκε και προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ από την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και ολόκληρη την Επιτροπή και όλος ιδιαίτερα σε την εισηγήτρια καθώς και όλους που προετοιμάσατε αυτές τις τροπολογίες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι στην Κομισιόν που βλέπουμε ισχυρή στήριξη για τους κεντρικούς στόχους της πρότασής μας και υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα μέτρα που προετοιμάζονται σε αυτό, με αυτό το κείμενο. Η αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά και να ε, επιτύχουμε λοιπόν τους ε, γενικούς μας ε, στόχους αλλά και τους ειδικούς μας στόχους. Οι τέσσερις ε, ήταν αυτοί. Πρώτος, επέκταση του πεδίου εφαρμογής. Θα ήθελα να σας πω ότι οι τροπολογίες είναι πολύ επικοδομητικές για το ζήτημα του ποιοι δρόμοι σε ποιου δρόμου θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Πολύ λίγοι από εσά αφισβητείτε την προτινόμενη επέκταση προ του 13 ε, κύριους δρόμους. Το να επεκτείνουμε μόνο στους αυτοκινητοδρόμους δεν αρκεί κατά τη γνώμη μας όσον αφορά τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα και τα ατυχήματα. Εμείς στόχο έχουμε το μηδέν τα μηδενικά ατυχήματα. Επίσης, κάποιες προτινόμενες προτάσεις ξεπερνούν την πρότασή μας γιατί περιλαμβάνουν ε, δρόμους της υπαίθρου και κύριους δρόμους. Ε, καλωσορίζω την προσπάθεια να, να υψώσετε τον πύχη ε, περισσότερο, όμως κάποιες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα φορτικές και βεβαρημένες και πιστεύουμε πως θα προκαλέσουν δυσκολίες ιδιαίτερα για τις τοπικές αρχές, επιπλέον βέβαια του κόστους, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να το σκεφτόμαστε και να είναι αναλογικό. Το δημόσια συζήτηση ίσως θα μπορούσε να μας διευκολύνει να, στην ε, τροπολογία 127 να ε, διευκρινίσουμε το κόστος. Ε, το θέμα του πεδίου εφαρμογή θα εξακολουθήσει να είναι σημαντικό για τη συζήτηση και στο τριμερή όπου γίνεται και σχετική συζήτηση εξάλλου στο Συμβούλιο. Στόχος από την πλευρά της Επιτροπής είναι να πούμε ξεκάθαρα ποια θα ήταν η επέκταση του πεδίου εφαρμογής που θα μας βοηθήσει να φτάσουμε σε όσο δυνατόν καλύτερη εφαρμογή. Έπειτα, ε, σηματοδότηση και ε, ε, σήμανση των δρόμων ε, είναι θέμα συνέπειας και συνοχής ανάμεσα στις δύο ε, προτάσεις για την οδική ασφάλεια. Από τη μια πλευρά έχουμε την, τον κανονισμό για την ασφάλεια των ε, οχημάτων και εδώ έχουμε την πλευρά των υποδομών και οι δυο αυτές νομοθεσίες θα πρέπει να συμβαδίσουν. Θα πρέπει δηλαδή το όχημα αλλά και ο δρόμος να μπορούν να έχουν επαφή μεταξύ τους και να προλαμβάνουν τα ε, λάθη και τα ανθρώπινα ακόμη λάθη. Τα αυτόνομα διοχήματα δεν λειτουργούν αν οι υποδομές δεν είναι έτοιμες. Σε διάφορες φάσεις αυτοματοποίησης θα είναι πολύ σημαντική επίσης η σηματοδότηση. Τρίτο στοιχείο της πρότασής μας είναι η αξιολόγηση του ε, δικτύου. Ε, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι μια διαδικασία με πραγματική συνέχεια ήταν μια από τις αδυναμίες που εντοπίσαμε στην ισχύουσα νομοθεσία του, δηλαδή οι διαδικασίες δεν ξέρουμε πώς ε, ακολουθούνται και αν οδηγούν σε δράση. Μπορεί να υπάρχει συνέχεια, να δίδεται συνέχεια, αλλά μπορεί και όχι. Και απλώ εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι που θέλουμε να διευκρινίσουμε με την, και με την 152, ότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συνέχεια και αυτό θα είναι πια υποχρέωση. Τέταρτος στόχο αφορά τους ευάλωτου χρήστες των δρόμων και αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για τους πεζούς, τους ποδηλάτε και τους μοτοσυκλετιστέ. Ανάλογα με το δρόμο βέβαια θα επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρονται εδώ ρητά για το είδος των δρόμων που εμείς έχουμε υπόψη μα. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που ζητούν από την Κομισιό να προχωρήσει περισσότερο. Για παράδειγμα, έχουμε μία για κοινά ε, μαθήματα για την ε, ε, μαθήματα οδήγησης και κοινέ εξετάσεις για τα διπλώματα. Θα είναι ενδιαφέρον να διερευνήσουμε και αυτές τις δυνατότητες, να αναπτύξουμε και ειδικά ειδικές απαιτήσει για τις υποδομές ε, για τους πεζούς, τις υποδομές για τα ποδήλατα, καθώς και κοινή μεθοδολογία για τα εθνικά σχέδια ασφάλειας. Όταν θα έχουμε φτιάξει τις ε, ειδικέ ομάδες ε, θα το, θα το προσεγγίσουμε και αυτό. Και για να κλείσω μια Ιδέα για το χρονοδιάγραμμα. Το Συμβούλιο θέλει να υιοθετήσει μια γενική προσέγγιση στις 3 ε, Δεκεμβρίου. Ελπίζω όλα να πάνε καλά στην Κορεπέρα αυτή τη βδομάδα. Πάντως η πρόθεση είναι αυτή. Πάντως η, πρόθεση αυτή, η πρόταση αυτή θα είναι ένα από τα θέματα που θέλουμε να ολοκληρωθούν μέσα σε αυτή τη θητεία. Εξαρτάται βέβαια αν μετά εσείς θα το υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Βερνά. Θα σας δώσω το λόγο κυρία Αγιούτο. Δύο λεφτά έχετε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπαν. Ε, προφανώς είναι και πολύ πιο θετικά όσον αφορά στο κείμενο και στις τροπολογίες, αλλά λιγότερο θετικά όσον αφορά σε ανησυχίες που εκφράζονται. Ε, Παραδείγματος χάρη αυτό που γίνεται σχετικά με την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξη, αλλά είμαι σίγουρη ότι τελικά θα κατορθώσουμε να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό, γιατί από τη μία πλευρά είναι ε, σημαντικό να ε, εξετάσει κανείς το θέμα του άχθους όσον αφορά στα κράτη-μέλη, αλλά όπως είπε και η Επιτροπή, αν ο στόχος μας είναι τελικά να περιορίσουμε ε, καθοριστικά τον αριθμό των θυμάτων, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν μέσα από την διεύρυνση. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι αυτή η διεύνηση και με ποιο τρόπο να λάβει η χώρα. Κατά τα άλλα θα συναντηθούμε την ε, Τετάρτη στη συνεδρία των σκιωδών εισηγητών. 3 Δεκεμβρίου θα είναι η ψηφοφορία. Αν χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ό,τι κατάλαβα, μπορείτε να μου στείλετε ένα mail για να την αναβάλουμε για αργότερη ψηφοφορία, για να υπάρχει έτσι μεταξύ και θέση του Συμβουλίου και να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Ωραία. Sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil. Πρόταση οδηγία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την τροποποίηση τη οδηγία 2106 για τα ελάχιστα πρότυπα κατάρτισης ε, των ναυτικών και για την κατάργηση της ε, Οδηγίας 45-2005. Δεν είναι εδώ ο εισηγητής, οπότε το λόγο έχει ο κύριος Τέλιτσκα. Ναι, τώρα δεν είμαι ο Βαν Μίλτεμπρουκ, είμαι ο Ντομερίκ Ρικέ. Σίγουρα πάντως δεν είμαι ο κύριος Κράμερ. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Έφυγε κιόλας. Anyway, uh, Uh, uh, λοιπόν, να επισημάνω ορισμένες παρατηρήσεις που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί σου ο Ντομινίκ. Χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την απλούστευση ε, και ενοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου για την επιγραμμική διαπίστευση των ε, ναυτικών και την ευθυγράμμιση των ε, ευρωπαϊκών προτύπων ε, με το διεθνή πρότυπα του IMO. Είναι κάτι το απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ποιοτική κατάρτιση των ναυτικών ε, που εργάζονται σε σκάφη, στην ευρωπαϊκή επικράτεια, αλλά και να παρακολουθούμε την ποιότητα των ναυτικών ε, που προσλαμβάνονται σε τρίτες χώρες. και σε παρελθόν αυτό είναι πρόβλημα. Και γενικά να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στα σκάφη. Επομένω, είναι θετική η διαδικασία αναθεώρηση ε, τη διαδικασία για τα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από τρίτε χώρε, από εκδίδονται από τρίτε χώρε και για την απόσυρση τη αναγνώριση. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ε, έχει δύο πλεύρε αυτό το νόμισμα. θα πρέπει να υπάρξει παράταση από τα 5 στα 8 χρόνια για την περίοδο απόσυρσης όταν δεν έχει υπάρξει πρόσληψη ναυτικών από τρίτες χώρε να εργαστούν σε σκάφος με ευρωπαϊκή σημαία. Αυτή η διευρυμένη περίοδος έχει ως στόχο να ακολουθήσει την διάρκεια κατάρτισης και διαπίστευσης. Από την άλλη, ο συγκητής θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη η πρόταση και προτείνει νέα μέτρα για τη βελτίωση της κατάρτισης για τους Ευρωπαίους ναυτικούς. Προτείνει λοιπόν ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αριστείας για τους ναυτικούς ε, που υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα ε, του διεθνούς δικαίου για να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και ε, να ευθυγραμμίσουμε τα προσόντα των ναυτικών με την ψηφιοποίηση των θέσεων εργασίας για να έχουν έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και μετά προτείνει τα πιστοποιητικά που εκδίδουν τα κράτη-μέλη ή αναγνωρίζονται από τέτοιες χώρες να μεταφέρονται σε βάση δεδομένων, αυτομάτως μάλιστα, σε κεντρική ε, ψηφιακή βάση δεδομένων. Με βάση και την οδηγία 16 του 2009 για το ε, κράτος λιμένα για να εξοικονομήσουμε ανθρώπινους ε, και οικονομικούς πόρους, να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος ε, εποπτείας συνολικά. Επιθυμεί να συνεργαστεί με τους σκιώδεις και να ξεβρεθεί συμφωνία πριν από το τέλος της θητείας. Δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσω αλλά είναι εδώ η ομάδα του Ντομινίκ και θα μεταφέρει ό,τι έχετε να πείτε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τέλσκα. Κύριε Μαρινέσκου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση. Νομίζω πως η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή και ότι η έκθεση του κυρίου Ντομινίκ Ρικέ είναι καλή. Κεντρική βάση δεδομένων και καλύτερη κατάρτιση για τους ναυτικούς. Θα ελέγξω αν πρέπει να καταθέσουμε περισσότερες τροπολογίες, αλλά για την ώρα πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσον. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιες ε, καλά σημεία στην έκθεση του κ. Ρικέ και, τα, ε, και είναι ευπρόσδεκτα ιδιαίτερα. Ε, συμφωνούμε με τον κύριο Τελίτσκα ότι η μετακίνηση προς ηλεκτρονικά συστήματα είναι θετική και αυτό το στηρίζουμε. Επίσης είμαστε πολύ ευτυχείς για την αναφορά στο πιστοποιητικό αριστείας ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η ε, το εργατικό δυναμικό των ναυτικών, ειδικά για τους αξιωματικούς, να είναι καλό ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκά αναγνωρισμένα τα προσόντα. Αυτό που δεν είπε όμως είναι ότι δυστυχώς αυτό μόνο αναφέρεται στα ε, εκτιμώντας. Και θα πρέπει να το σοβαρά να το σκεφτούμε, όπως ε, ας πούμε για τα λιμάνια όταν κάναμε ε, την σχετική οδηγία πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό άρθρο και να μπει στο διατακτικό. Θα το συζητούσαμε τον κύριο Τέιλορ και τον κύριο Μαρινέσκο αυτό. Ε, είναι καλή αρχή δηλαδή, αλλά λίγο περισσότερη δουλειά χρειάζεται. Επίσης ένα πιθανό πρόβλημα και ίσως αυτό να οφείλεται σε δική μου παρεξήγηση είναι ότι η τροπολογία 10 του κυρίου Ρικέ αφαιρεί την αναφορά και υπογραμμίζει τη σημασία των περιόδων ανάπαυσης στις 3 ώρες. Είμαι βέβαιος ότι δεν, ε, βέβαια ότι δεν έχει την ε, πρόθεση να απομακρυνθεί από ε, τις θεσμισμένες ώρες εργασίας των ναυτικών. Ίσως θα πρέπει να γίνει λοιπόν κάποια διευκρίνηση γιατί μπορεί έτσι να δημιουργηθούν προβλήματα. Θα θέλαμε λοιπόν αυτό να επανεξεταστεί. Και έπειτα υπάρχουν και διάφορα ζητήματα ε, αναγνώρισης τρίτων χωρών ε, για στόχους ε, των ναυτικών. Ας πούμε, αναγνώριση χωρών που δεν έχουν εκπαιδεύσει ναυτικούς εδώ και χρόνια. Αυτό είναι πρόβλημα όσον αφορά την αυτόματη αναγνώριση στο Συμβούλιο. Τα 8 χρόνια νομίζω δεν είναι ο καλύτερος τρόπος, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ποια χρονική περίοδος για χώρες που δεν έχουν ε, προσφέρει στην Ένωση ναυτικούς, αναγνωρισμένους ναυτικούς, τότε η αναγνώριση αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε όλα τα συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί να προκέψουν. Δεν είμαι πεπισμένο λοιπόν για το, για το 5, το 8 και το 7. ως σκιώδης θα πρέπει να κάνουμε μια γνήσια συζήτηση για όλα αυτά και ξέρω σε κάποιο βαθμό υπάρχει πίεση να ξεμπερδέψουμε με για την υπόθεση αλλά ελπίζω πως θα έχουμε πραγματικά χρόνο να εξετάσουμε αυτά τα θέματα γιατί είναι σοβαρά. Και έπειτα παρόμοιο θέμα για την αναγνώριση των μεμονωμένων πιστοποιητικών ναυτικών από τρίτες χώρες. Ε, χρόνος που χρειάζεται να υπάρχει ώστε να εξασφαλίσουμε ότι εξετάζονται αυτά τα πιστοποιητικά και ότι η έμσα που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι υπερφορτωμένη ή υπερχαλαρή. Άρα λοιπόν και εκεί θα πρέπει κάπως να το σκεφτούμε. Εκ πρώτης είναι απλή λοιπόν η πρόταση αυτή και ναι, ξέρω πάντοτε το λέω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει στην πράξη υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν πιο ενδελεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Άντερσον. Κύριε Τέιλορ, έχετε τώρα εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ στον κύριο Χικέ που λείπει. Η πράσινη, λοιπόν ε, μπορούν να στηρίξουν πάρα πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνει το κείμενο και συμφωνούμε και με το ότι εκφράζεται ανησυχία ε, σχετικά ε, με την ασφάλεια αυτών των ναυτικών. Πράγματι, να υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό αριστείας ε, το οποίο να ξεπερνάει τις ελάχιστες προδιαγραφές, όπως επίσης ε, και την ιδέα να υπάρχει μια κεντρική τράπεζα δεδομένων για τα πιστοποιητικά που εκδίδουν τα κράτη-μέλη. Για να προσόφελος των σκαφών και των πληρωμάτων είναι επιγόντως απαραίτητο να ελέγχεται η ποιότητα της εκπαίδευσης των ναυτικών συμπεριλαμβανομένης και της ποιότητας εκπαίδευσης εκείνων που έχουν προσληφθεί σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ρυθμίσεις για την αναγνώριση των πιστοποιητικών από τις τρίτες χώρες και η αμοιβαία αναγνώριση ε, των ε, πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα κράτη-μέλη, όλα αυτά να είναι ε, επαρκώς διαφανή και δίκαια. Ευχαριστούμε. Στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνω το λόγο στην κυρία Κοψίνσκα. Τι γίνεται το πόδι, καλά? Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ που ρωτάτε για το πόδι μου ε, ε, Σαφώ και πάει καλύτερα. Πάντα όταν έρχομαι στο κοινοβούλιο πάνε όλα καλύτερα όσον αφορά στην υγεία μου. Ε, τώρα, όσον αφορά τον εισηγητή, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή αλλά και του ε, σκιώδει εισηγητέ ε, για τη δουλειά του, για τα σχόλιά του. Ξεκινώντα, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ επικοδομητικό αν τελικά Είχαμε μια σύντομη συνάντηση με τον εισηγητή και τους και εισηγητές για να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που ετέθησαν εδώ, γιατί νομίζω ότι συμφωνούν όλοι ότι συμφωνούν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ίσως να διαφωνούν με κάποια διατύπωση που ενδεχομένως να οδήγησε σε κάποια παρεξήγηση και σε επίπεδο εισηγητή και όσον αφορά τις ε, ερωτήσεις σας. Ε, χαίρομαι που ο εισηγητής ε, διατηρεί την φιλοδοξία τη δική μας έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί το δικό μας το σύστημα με την σύμβαση SDWC για να είμαστε σίγουροι ότι διασφαλίζεται ένα επίπεδο εκπαίδευση όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άλλα σκάφη ε, που δεν είναι ευρωπαϊκά ή ενωσιακά, έχουν όμως ενδεχομένως ε, την ευρωπαϊκή σημαία. Επίσης, χαιρόμαστε και για την πρόταση να ασκηθεί πίεση για την ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών για τους ναυτικούς. Καλή και πρόταση για κεντρική τράπεζα δεδομένων των πιστοποιητικών να συσταθεί αυτή το συντομότερο δυνατόν. Όπως σας είπα, υπάρχουν κάποια θέματα που τίγονται στην έκθεση και κατά την την άποψή μου οδηγούν σε παρεξήγηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρόταση επέκτασης από 5 σε 8 έτη η περίοδος κατά την οποία στο τέλος ε, θα μπορεί να υπάρχει αναγνώριση. Ξέρετε, αυτή δεν είναι αυτόματη η απόσυρση. Ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια απόφαση για να υπάρξει απόσυρση και τα πέντε χρόνια έχουν σχέση με την διάρκεια ισχύω ε, ε, του πιστοποιητικού ικανότητας άρα σας λέω το πέντε δεν, είναι, δεν το διαλέξαμε τυχαία η όλη ιδέα είναι ότι θέλουμε να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τους πόρους ε, της ΕΜΣΑ που πρέπει να διατίθενται για επιθεωρήσεις αν τελικά δεν δεν υπάρχει κανένα ναυτικός ε, που να έρχεται από τη χώρα για την οποία έχει ζητηθεί η αναγνώριση. Απλά ε, είναι η αναγνώριση της δουλειάς που πρέπει να κάνει η ΕΜΣΑ. Επίσης, Συμφωνώ αυτά που ελέγχθηκαν, ελέγχθησαν σχετικά με την τροπολογία υπαριθμών 10, το ελάχιστο της ανάπαυσης. Το να αφαιρέσουμε αυτό είναι απλά μία παρεξήγηση, αλλά παράλληλα θέλω να σας πω όπως είπα και στην αρχή, ότι η πρόταση ζητά την ε, ψηφιοποίηση όλων των πιστοποιητικών για τους ναυτικούς. Αυτό εμείς ε, το χαιρετίζουμε και πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που χρήζει διευκρίνησης είναι η όλη διαδικασία ε, της αναγνώρισης. Δεν είναι μια διαδικασία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτίθεται να κάνει κάτι μόνη της. Έχουμε μια διαδικασία που ισχύει σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Έχουμε μια συζήτηση με τα κράτη-μέλη για το κατά πόσον θα πρέπει να προχωρήσει η αναγνώριση. Γιατί μερικές φορές βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ένα κράτος μέλος μας ε, γράφει και λέει παρακαλώ αναγνωρίστε το κράτος Χ ε, δεν είναι λοιπόν μια ιδέα την οποία υποστηρίζουν όλοι οι επιφύλακτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω εκ τούτου το να συζητηθεί αυτό στην Επιτροπή έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και με όλα τα κρατημέλη και όχι μόνο με εκείνα που ζητούν την αναγνώριση. Πέρα από αυτό νομίζω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς ε, η ολοκλήρωση της έκθεσης ε, θα μας οδηγήσουν σε μια πολύ καλή πρόταση. Το Συμβούλιο ελπίζω να είναι έτοιμο να δεχτεί την ευρύτερη προσέγγιση. Πιστεύω ότι τελικά θα μπορέσουμε ε, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το νομοθέτημα σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπενθυμίζω ότι τροπολογίες μπορείτε να καταθέσετε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Τα ξαναλέμε αύριο στις 9 το πρωί, όπου έχουμε μια πολύ μεγάλη ψηφοφορία, γιατί ξεκινούμε από το ΣΕΦ. Έτσι δεν είναι κύριε Μαρινέσκου τα ξαναπούμε αύριο στις 9. Et à demain, merci à vous. Merci les traducteurs. Euh, non, les interprètes, excusez-moi. Η Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τους δερμηνείς. Καλό σας βράδυ.